Καλησπέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Είμαστε λίγοι, αλλά ελπίζω να γίνουμε περισσότεροι. Πάντα είναι δύσκολα τα πράγματα τις Δευτέρες το απόγευμα. Ήδη αφήσαμε ένα δεκάλεπτο για να προλάβουν να έρθουν οι συνάδελφοι. Τώρα δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο. Καταρχήν, ε, ο πρόεδρο ζητά συγγνώμη για την απουσία του. Ο, ο κύριο και ο πρόεδρό μα κολλείται για σήμερα το απόγευμα. Και γι' αυτό τον αντικαθιστώ εγώ στην Προεδρία. Επίσης, να ξεκινήσουμε με τα σημεία της ημερήσιας διάταξης. Καταρχήν, έγκριση της, ε, του σχέδιου ημερήσιας διάταξης. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσει για το προτινόμενο πρόγραμμα, θεωρώ ότι εγκρίνεται η μερίσια διάταξή μας. Σημείο 2. Ανακοινώσεις ε, της Προεδρίας. Το μόνο που έχω να σας πω είναι ότι ως συνήθως και η σημερινή μας συνεδρίαση θα μεταδοθεί στο διαδίκτυο από το web streaming. Και παρόλο που είμαστε λίγοι, θα σας υπενθυμίσω, θα το παραλάβω και αργότερα, ότι κατά το τέλος της συνεδρίασης, στις 7 δηλαδή το απόγευμα, στην ίδια αίθουσα θα παραθέσουμε μια μικρή δεξίωση χριστουγεννιάτικη. Οπότε μετά το πέρας των εργασιών. Στις 7 η ώρα είστε όλοι καλεσμένοι στο κοκτέιλ που θα οργανώσουμε ένα Χριστουγέννων. Στην ίδια αίθουσα επαναλαμβάνω στις 7. Θα το επαναλάβω και αργότερα γιατί λίγοι συνάδελφοι είναι παρόντες για να ενημερωθούν όλοι για τη μικρή αυτή δεξίωση. Επίσης, μην ξεχνάτε ότι προβλέπεται διερμηνία σε 18 γλώσσες με εξαίρεση τα τσεχικά, λετωνικά, μαλτέζικα, σλοβακικά, ε, δανέζικα και γοεδελικά. Συγγνώμη, δανέζικη διερμηνία προβλέπεται. Ε, Επίσης, έγκριση των πρακτικών της 5 η Νοεμβρίου του 2018. Αν δεν υποβληθούν παρατηρήσεις ή αντιρρήσεις μέχρι το τέλος της συνεδρίασης, θα θεωρηθούν ως συγκεκριμένα. Και περνάμε στο σημείο 4. Παρουσίαση της έκθεσης σχετικά με την αποστολή της Επιτροπής Άγκρης στη Βουλγαρία που πραγματοποιήθηκε 29 με 31 Οκτωβρίου. Ήταν η τελευταία μας αποστολή. 29 με 31 Οκτωβρίου 2018 στη Βουλγαρία. Μια αντιπροσωπεία της Επιτροπής Γεωργίας επισκέφθηκε εκείνες τις μέρες στη Βουλγαρία. Ο Μόμτσιλ Νέκοφ των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών από τη Βουλγαρική Αντιπροσωπεία, οργάνωσε μαζί με τον Βλαντιμίρ Ούρουτσεφ από το ΕΛΚ τη σχετική αποστολή. Στην αποστολή συμμετείχαν ο πρόεδρος Εκέρσκι, ο κύριος Ντόρφαν, η Μαρία Νόιχλ, ο Μάρκ Ταραμπέλα, η Λίδια Σένρα Ροδρίγκες και ο Ζακ Κολομπιέ. Στόχος της αποστολής ήταν η αξιολόγηση των επιτυχιών και των προκλήσεων της ε, πρόσφατης βουλγαρικής προεδρίας στα θέματα της γεωργίας. Και εγώ ως ε, εισηγήτρια για τις φαρμακούχες ζωοτροφές θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμότατα την ε, Βουλγαρική Προεδρία για τις προσπάθειες που έκανε στα θέματα της υγείας των ζώων. Το επίσημο πρόγραμμα περιλάμβανε κάποιες θεσμικές συναντήσεις με τον Βούλγαρο Υπουργό Γεωργίας και το επιτελείο του, με την πρόεδρο της Επιτροπής Γεωργίας της Βουλγαρικής Βουλής, συναντήσεις με μη κυβερνητικές οργανώσεις και εκπροσώπους ε, γεωργών, καθώς και επισκέψεις ε, σε πολλές αγροτικές περιοχές. Τα μέλη της αντιπροσωπείας είχαν μια πραγματική γνήσια ε, βουλγαρική εμπειρία και μάλιστα με ηλιόλουστο κλίμα, από ό,τι μου είπαν. Οπότε και ο καιρός βοήθησε. Θα μας το εξηγήσετε σε λίγο. Έχουμε μάλιστα μια διεξοδική έκθεση από τη γραμματεία για τα πεπραγμένα της αποστολής που σας τη στείλαμε και ηλεκτρονικά. Πριν λοιπόν περάσουμε στη συζήτηση θα ήθελα να ευχαριστήσω εκ μέρους της Επιτροπής μας τους κυρίους Νέκοφ και Ουρουτσέφ για την διοργάνωση αυτή της αποστολής και για το πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα που εκπώνησαν. Ο κύριος Νέκοφ απουσιάζει από ό,τι βλέπω. Δεν ξέρω, είναι παρόν ο κύριος Σούρουτσεφ ε, για να μας ενημερώσει. Παρακαλώ. Μπορείτε να μας ε, πείτε δύο λόγια για την αποστολή και την εμπειρία που αποκομίσατε σε αυτή την επίσκεψη στη Βουλγαρία. Κύριε Ρουτσέφ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι. Πολύ ευχαριστώ να σας παρουσιάσω τα τελευταία αποτελέσματα της ε, Επιτροπής μας στα τέλη Οκτωβρίου της αποστολής στην Βουλγαρία με 8 βουλευτές η ομάδα μας από 4 πολιτικές ομάδες και καταρχάς θα ήθελα να επισημάνω ότι πρόκειται για την πρώτη επίσημη αποστολή της Επιτροπής μας στη Βουλγαρία, ύστερα από την προσχώρηση της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία οργανώθηκε μήνες μόλις μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των εργασιών της ε, Βουλγαρικής Προεδρίας του Συμβουλίου που επεξεργάστηκε τα θέματα της ΚΑΠ μετά το 2020. Στόχος αυτής της τρίμερης επίσκεψης ήταν μια στενότερη επισκόπηση των ε, μέχρι τώρα εμπειριών αλλά και των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι αρχές της Βουλγαρίας και οι διάφοροι φορείς που έχουν να κάνουν με την υλοποίηση της κοινή γεωργικής πολιτικής αλλά και η παρουσίαση από πλευράς τους ε, των προτάσεών τους για την περίοδο μετά το 2020. Για την κάπου μετά το 2020. Είχαμε συνεδριάσεις με τον Υπουργό Γεωργίας, με εκπροσώπους του Υπουργείου, των κλάδων Γεωργίας ε, Τροφίμων Δασοκομείας Γενικό ε, Πρόεδρο της Επιτροπής ε, Γεωργίας της Βουλής της Βουλγαρίας αλλά και μέλη της Επιτροπής αυτής και συνεδρίαση με μη κυβερνητικέ οργανώσεις του γεωργικού κλάδου. Είχαμε πάνω από 15 οργανώσεις που εκπροσωπούν μια σειρά από τομείς, τομέα ε, δημητριακών, προκυπευτικών, κτηνοτροφίας, βιολογικής γεωργίας, νεαρούς, ε, γεωργούς και άλλους. Ε, επισκεφθήκαμε επίσης ε, κέντρα ε, διήλυσης για το ροδέλαιο, άλλες εγκαταστάσεις, ινοπαραγωγούς. Συζητήσαμε προτάσεις για το μέλλον της ΚΑΠ και την ε, προσαρμογή στις ε, εθνικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες, της ε, προσαρμογή της ΚΑΠ στις ιδιαιτερότητες της Βουλγαρίας και τις ανάγκες της. Όλοι μίλησαν μια καλύτερη χρηματοδότηση της ΚΑΠ και απλουστευμένες διαδικασίες για τους δικαιούχους. Τα νότατα επίπεδα των άμεσων ενισχύσεων το μοντέλο άμεσης ε, αποτελεσματικότητας ή πρόσβαση στη γεωργική γη για νέους γεωργούς που μάλιστα οδήγησε σε έντονες αντιπαραθέσεις απόψεων. Γιατί υπάρχει νέα νομοθεσία που ετοιμάζεται στη Βουλγαρία αυτή τη στιγμή η οποία θα διευκολύνει την πρόσβαση στην αρρώσιμη γη για τους γεωργούς Ιδιαίτερη προσοχή επίσης δόθηκε στην πρόσθετη υποστήριξη του τομέα των βοηδών, ρηστευρωμένες ε, ενισχύσεις σε τομείς ευαίσθητους όπως η των του καπνού, που αποτελεί σημαντικό πόρο και πηγή βιοπορισμού για ορισμένες περιοχές απομακρυσμένες και ορεινές. Και καταλήγοντας, θα ήθελα να πω πως ε, θεωρούμε επικοδομητική και παραγωγική την επίσκεψη. Ήταν πολύ καλή η οργάνωση, η ποιότητα των συζητήσεων, η επισκέψεις. Τα μέλη της Επιτροπής μας μπορέσαν να δουν η διεισόμαση ότι υπάρχει μεγάλο δυναμικό με μοναδικά προϊόντα, προϊόντα υψηλής ε, ποιότητας και βέβαια ότι η γεωργία έχει κέριο χαρακτήρα για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριο Ρούτσεφ. Το λόγο έχει τώρα ο κύριος Ταραμπέλα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν θα είμαι πιο αναλυτικός από τον συνάδελφο που μας υποδέχτηκε στη Βουλγαρία γιατί στην πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η αποστολή, όχι μόνο για μένα, για όλους τους συναδέλφους, γιατί ανακαλύψαμε την γεωργική πτυχή της Βουλγαρίας. Είδαμε ότι είναι μια πολυλειτουργική γεωργία. Έχουμε ε, σιτοπαραγωγή, κτηνοτροφία, ε, προβατοτροφία και μάλιστα πριν από μερικά χρόνια είχαμε 16 εκατομμύρια, τώρα έχουν μείνει πολύ λιγότερα εκατομμύρια προβάτων, ενώ εισάγουμε από την άλλη άκρη του πλανήτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρόβιο κρέας. Πολύ ενδιαφέρουσα ήταν πάντως αυτή η επίσκεψη. Ε, μάλιστα συναντήκαμε και την Υφυπουργό Γεωργία, την κυρία Κράστεβα και με πολλές μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Και δεν θα σας το γεγονός ότι η παραγωγή δημητριακών είναι κατά του κάπινγκ των ενισχύσεων, ενώ οι κτηνοτρόφοι κρίνουν σκόπιμο κάτι τέτοιο. Γιατί ξέρουν ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ενισχύσεων ωφελεί μια μικρή μονομάδα παραγωγών. Επίσης, ε, επισκεφτήκαμε και μια βιολογική γεωργική εκμετάλλευση που και στη, σε υπαίθρια καλλιέργεια αλλά και σε θερμοκήπιο είχαμε εκτεταμένη παραγωγή απορροκυπευτικό και κυρίως ε, οσπρίων, ψυχανθών. Επίσης ε, είχαμε στην ε, Δαμασένα όπου ένα εκτάριο ε, ροδοκαλλιέργειας ε, είχαμε παρήγαγε ένα, ένα, ένα, ε, ένα λίτρο χρειάζονται 9 τόνοι, για να παραχθεί, 9 τόνοι ροδοπετάλο για να παραχθεί ένα λίτρο, 30, ένα λίτρο ροδέλαιο. είναι τεράστιο το έργο δηλαδή που χρειάζεται για να παραχθεί το ροδέλαιο. Επίσης είχαμε ε, και συνάντηση με μελισσοκόμους εδώ στις Βρυξέλλες ε, ε, επί ε, θητείας κυρίας ε, Γκαμπριέλ. Τότε είχε ετοιμάσει αυτή την επίσκεψη των μελισσοκόμων εδώ και, και εκεί στην Καλοφέρη είδαμε ποια είναι τα δυνατά σημεία της βουλγαρικής μελισσοκομείας και ποιες είναι οι προσδοκίες των Βουλγάρων και άλλων μελισσοκόμων. Επίσης, ε, πήγαμε, περάσαμε από το Πλόφτη, δεν σταματήσαμε εκεί, αλλά ε, ε, είχαμε το Μαυρούδι που είναι μια τοπική ποικιλία. Ήταν αδύνατο να πάμε στη Βουλγαρία χωρίς να επισκεφτούμε αμπελουργίες στον αμπελονικό κλάδο. Και επίσης την τελευταία μέρα επισκεφθήκαμε την Βουλγαρική Βουλή και μας υποδέχθηκε η κυρία Καριάντσεβα, η πρόεδρος της Βουλής και η πρόεδρος Τη Επιτροπή Γεωργίας τη Βουλή. Κυρία Τάνεβα, είχαμε μια πολύ επικοδομητική συζήτηση με του συναδέλφου και εκεί συζητήσαμε τα, τις προτάσεις μεταρρύθμισης ε, με κοινού φόβου που έχουν και οι Βουλγαροί για τη Γεωργία και την κοινή γεωργική πολιτική. Πάντως, πολύ, ήταν, πολύ επικοδομητική ήταν αυτή η αποστολή στη Βουλγαρία και ευχαριστώ του συναδέλφου Νέκοφ και Ουρουτσέφ για το άρτιο, πολύ πυκνό πρόγραμμα, πολύ ισορροπημένο, γιατί είχαμε ταυτόχρονα και επίσημε συνεδριάσει αλλά και επισκέψει επιτόπου. Εκεί συλλέξαμε πολύ χρήσιμε πληροφορίε που θα μα εμπνεύσουν και στο μέλλον στι συζητήσει. Ευχαριστώ, Μάρκ. Θα ήθελα να καλωσορίσω κάποιους ε, νέους φοιτητές από το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελών μετά από πρόσκληση του Παύλου Ντεκάστρο Καλώς ήρθατε. Αν δεν κάνω λάθος και εσείς ασχολείστε με την κοινή γεωργική πολιτική και ελπίζω η εμπειρία εδώ στην Επιτροπή Γεωργίας να σας ε, χρησιμεύσει. Ο κυρία Νόιχλ έχει το λόγο. Θα ήθελα επί ευκαιρία να ευχαριστήσω το προσωπικό μας, γιατί ένα τέτοιο πρόγραμμα δεν ε, πέφτει από τα δέντρα, ε, κρύβει πίσω του πάρα πολύ δουλειά ήταν πάρα πολύ καλά οργανωμένη άρτια αυτή η επίσκεψη και θέλω να ευχαριστήσω ρητά. Θα ήθελα λοιπόν να εστιαστώ στα εξή δύο. Συγκέντρωση γεωργικής γη. Εάν 6% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων εισπράττουν το 90% των επιδοτήσεων στη Βουλγαρία, τότε νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα να ξανακοιτάξουμε το πώ θα γίνει η αναδιανομή των ενισχύσεων. Οπωσδήποτε η κατανομή των, των ενισχύσεων με βάση την έκταση τη γεωργική αποδεικνύεται άδικη. Και νομίζω ότι πρέπει να κοιτάξουμε ποιε είναι εκείνε οι επιχειρήσει οι οποίε είναι στραμμένε προ το μέλλον, είναι ανοιχτέ προ τι εξελίξει. Γιατί το έχουμε και αυτό και στην ε, Βαβαρία. Ακόμα και μεγάλε επιχειρήσει μπορεί να είναι στην πρωτοπορία, αλλά υπάρχουν και μικρέ ε, επιχειρήσει γεωργικέ με τρία-τέσσερα στρέμματα πίσω από το σπίτι, επί παραδείγματι, που και αυτές θα μπορούσαν να λαμβάνουν ενίσχυση. Έτσι λοιπόν, όταν έχουμε μια τέτοια μεγάλη, τόσο μεγάλα, μεγάλη διαφορά σε ένα κράτος όπως η Βουλγαρία, ε, με τα απορροκυπευτικά ιδιαίτερα που ε, είδαμε. Οπωσδήποτε δεν μπορεί να είναι στόχος Ευρωπαϊκής Ένωσης να ενισχύονται οι μεγάλες γεωργικές επιχειρήσεις ε, επειδή αποδυναμώνονται οι ανταγωνιστές τους, οι μικρότερες επιχειρήσεις. Ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει με την αναισθητοποίηση των ζώων. Ίσως θα θυμούνται, θα γνωρίζουν τα θέματα καλύτερα οι συναδελφοί. Είχαμε ένα ζήτημα με την ε, έκκληση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, την επικονίαση, η οποία έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Πρέπει να τιμηθεί ο μελισουργός που εξασφαλίζει την επικονίαση, χωρίς τον οποίο, χωρίς τη μελισουργία δεν θα μπορούσε να γίνεται η επικονίαση, η γονιμοποίηση και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το υποστηρίξουμε. Μπορεί να πει κανείς, μπα δεν είναι τίποτα. Όχι, νομίζω όμως ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία και το μέγεθος των επιχειρήσεων στην υπόθεση αυτή και θα πρέπει να το κοιτάξουμε όπως πρέπει να κοιτάξουμε και την μελισουργία και την επικονίαση με τον τομέα των οποροκυπευτικών που έχουν τεράστια σημασία. Εδώ πρέπει να βελτιώσουμε, να βελτιώσουμε τις επιδόσεις μας. Ξέρω ότι έχει περάσει η προθεσμία για την καταθέση των τροπολογιών για την κυριολογική πολιτική. Έχει περάσει πλέον ε, η προθεσμία, αλλά πρέπει ό,τι μπορούμε να κάνουμε για να στηρίξουμε την ε, Γεωργία στη Βουλγαρία ιδιαίτερω και όχι να επιτρέψουμε μέτρα τα οποία μπορεί να υποβούν βάρος της. Και πάλι ευχαριστώ για την οργάνωση. Κυρία Λίδια το λόγο. Ευχαριστώ. Ήταν πολύ καλή διοργάνωση, πολύ φιλόξενη υποδοχή. Δεν θα σας αναφέρω λεπτομεριακά τις επισκέψεις που πραγματοποιήσαμε, γιατί με κάλυψαν ε, οι προλαλήσαντες. Αυτό που εμένα μου έλειψε ήταν δύο επισκέψεις, δύο συναντήσεις. Μία με γυναίκες αγρότησες, γυναίκες της υπαίθρου των αγροτικών περιοχών, γιατί είχαμε πει και είχαμε συμφωνήσει ότι σε όλες μας τις επισκέψεις θα πρέπει να συναντούμε γυναίκε αγρότησες. Στην περίπτωση αυτή όμω δεν είχαμε τέτοια ευκαιρία. Και επίση ε, επισκέψει και συναντήσει με μικροκαλλιεργητέ, γιατί είδαμε κυρίω ε, μεγάλε έκταση αγροτικέ εκμεταλλεύσει. Κρίμα που δεν είχαμε επαφή ή συνάντηση με γεωργού, μικροκαλλιεργητέ ε, για γεωργία μικρή κλίμακο. Η υπόλοιπη επίσκεψη ήταν πολύ χρήσιμη, αλλά στο μέλλον αυτά τα δύο στοιχεία θα ήθελα να μην λείπουν από τα προγράμματά μα. Ευχαριστώ, Λίδια. Δεν ξέρω αν ο κύριος Σούρουτσεφ έχει να προσθέσει κάτι. Έχει το λόγο σύντομα, αν θέλει, αλλά δεν είναι υποχρεωμένο. Αν θέλετε το λόγο, ευχαρίστω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τους συναδέλφους για την πολύ ε, πιστή περιγραφή της αποστολής. Καταφέραμε όντως χάρη στις συναντήσεις που είχαμε να αντιληφθούμε τα πιο ζωτικά προβλήματα της βουλγαρικής γεωργίας και θα μας χρησιμεύσει όλη αυτή η εμπειρία. Ευχαριστώ για την υποστήριξή σας. Είναι προφανές ότι ελάχιστα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την ΚΑΠ για να επιλύσουμε κάποια βασικά προβλήματα της βουλγαρικής γεωργίας. Πάντως, σε εθνικό επίπεδο έχουμε επίγνωση των προβλημάτων και ήδη αναζητούμε λύσεις σε νομοθετικό επίπεδο στη χώρα. Ευχαριστώ και πάλι θερμά του συναδέλφου που έλαβα μέρο στην αποστολή αυτή και θεωρώ ότι πραγματικά στέφθηκε με επιτυχία. Ρουτσεφ. Ευχαριστώ κύριε Ρουτσεφ και όχι μόνο εσά και όλου του συμμετέχοντες, γιατί βλέπω ότι όντως ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η αποστολή στη Βουλγαρία. Ας περάσουμε τώρα στο σημείο 5 της ημέρησιας διάταξης. Προβλέπει παρουσίαση από εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της κατάστασης προόδου ό,τι αφορά τον κατεξιδότηση κανονισμό της Επιτροπής της 17 Οκτωβρίου του 2018 που συμπληρώνει τον κανονισμό 1308 κάθετος 2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με θέμα της αιτής προστασίας ονομασιών προέλευσης γεωγραφικών ενδείξεων και παραδοσιακών ενδείξεων στον αμπελονικό τομέα, τη διαδικασία ένστασης, τους περιορισμούς στη χρήση, τη τροποποίηση των προδιαγραφών προϊόντων, την ανάκληση της προστασίας, καθώς και την επισήμανση και την παρουσίαση. Στις 22 Φεβρουαρίου του 2018, η Επιτροπή μας ε, άκουσε την παρουσίαση του σχεδίου κατεξουδότηση πράξη από χετρία κεφάλαια. Τις προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης, τις γεωγραφικές ενδείξεις, τις παραδοσιακές ενδείξεις, την επισήμανση και την παρουσίαση. Όλα τα μέλη της Επιτροπής άκουσαν με ικανοποίηση την παρουσίαση της πρώτης Ευρωπαϊκής επιτροπή και την έκριναν ω ε, γνήσια ε, απλούστευση της κατάστασης στον κλάδο στα πλαίσια του ενιαίου ε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μάλιστα η κατεξοδότηση πράξη οθετήθηκε από την Επιτροπή και μεταβιβάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 17 Οκτωβρίου. Εξού και η προθεσμία για την υποβολή αντιρρήσεων ορίστηκε για την 17η Δεκεμβρίου του 2018. Και μάλιστα 5 ε, Νοεμβρίου του 2018 ήταν η εσωτερική προθεσμία της Επιτροπής μας για την η υποβολή αντιρρήσεων και τότε ο κύριος Δεκάστρο ζήτησε και επίσημα μια παράταση της ε, περίοδου διενέργειας ελέγχου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτής κατά εξοδότηση πράξης. Ο κύριος Δεκάστρο ε, στήριξε την ε, ανησυχία του στην αιτιολογική σκέψη 45 που σχετίζεται με το άρθρο 51 και αφορά τα προϊόντα του αμπελοϊνικού κλάδου που δεν καλύπτονται από προστατευόμενη ονομασία προέλευση ή γεωγραφική ένδειξη. Στις 21 Νοεμβρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαβίβασε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μια διόρθωση αυτής της κατεξοδότηση πράξης προκειμένου να διορθωθεί ένα σφάλμα που περιλαμβανόταν σε όλες τις μεταφράσεις ε, πλήν των αγγλικών ε, και γι' αυτό στην αιτιολογική σκέψη ο όρος ε, μετα... χώρα μεταποίησης αντικαταστάθηκε από τον όρο χώρα παραγωγής, το processed of the produced. Ο κύριος Δεκάστρο ζήτησε να συζητηθεί αυτό στην τελευταία συνεδρία των συντονιστών και να καλέσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για μια ανταλλαγή απόψεων για το θέμα αυτό. Αυτό ακριβώς κάνουμε σήμερα. Γι' αυτό και μετά από εντολή των συντονιστών διοργανώσαμε τη σημερινή συζήτηση για να ακούσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις εξηγήσει και την παρουσίαση της κατάστασης. Θα καλωσορίσω τον κύριο Ζωάο Νοφρέ της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας που είναι υπεύθυνος για το ζήτημα αυτό. Κύριε Νοφρέ, έχετε το λόγο. Alignment of the, σύμφωνα με τον κανονισμό 607 σε ό,τι αφορά τις γεωγραφικές ενδείξεις, την α, παρουσίαση και την επισήμανση, η πράξη κατεξουσιοδότηση υιοθετήθηκε από την Επιτροπή στις 16 Οκτωβρίου και η πράξη εφαρμογής θα α, α, υιοθετηθεί σε συνέχεια της συνάντησης αυτής. Τα τελευταία τρία χρόνια η Επιτροπή δούλεψε μαζί με τα κράτη-μέλη αλλά και εκπροσώπους του παρόντο τομέα, καταφέραμε να καταλάβουμε ο ένα τα συμφέροντα και τι ανησυχίε του άλλου και στο τέλο, η Επιτροπή ήταν πεπισμένη ότι στο τέλο της διαδικασία, όλα τα, μέλη, τα μέρη κατέληξαν να είναι ικανοποιημένα. Αυτό είναι μέρος ευθυγραμμισμού με τη συνθήκη τη Λισαβόνα, κάτι που έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πολύ καιρό επίγει και είναι πολύ σημαντικό για την ανάπτυξη του αμπελουργικού τομέα να έχουμε ένα νομικό πλαίσιο θα ήθελα να είμαι εξαιρετικά σαφής σχετικά με αυτήν την πράξη κατά εξουσιοδότηση και με το ότι δεν περιλαμβάνει. Κατά τη διάρκεια της περίοδου εξέτασης, ένα συγκεκριμένο λάθος που βρίσκεται σε μια αιτιολογική σκέψη διαβάστηκε ως εξής. σε ό,τι αφορά την επισήμανση των μη γεωγραφικών ενδείξεων, κάτι το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει σε παρεξηγήσεις. Η Επιτροπή άμεσα υιοθέτησε ένα διορθωτικό κείμενο, ούτω ώστε να μπορέσουν να αποτρέψουν οποιαδήποτε ανησυχία. Κατά συνέπεια, δεν υπάρχει καμία περίπτωση σε ό,τι αφορά τις επινσημάνσεις ίνου που προέρχεται μίας και μόνης ποικιλία να δημιουργηθεί παρεξήγηση η υποχρέωση να ονομάζεται η γεωγραφική ένδειξη παραμένει πιο σημαντικά. Τώρα, όπως και στο μέλλον, δεν υπάρχει πιθανότητα εισαγωγής, α, εισαγωγής κρασιών και σταφυλιών από κάποια άλλη χώρα και μουστου χωρίς να αναφέρεται η γεωγραφική προέλευση. Αυτό που θα ήθελα να τονίσω τώρα είναι τι περιλαμβάνει ο κανονισμός αυτός. Ε, υπάρχει μια πάρα πολύ σημαντική απλούστευση σε ό,τι αφορά τον ίνο μίας και μόνης ποικιλία και ιδίως σε ό,τι αφορά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Α, ο κανονισμός αυτός ευθυγραμμίζεται με κανονισμούς για άλλα προϊόντα και τρόφιμα και μπορεί να εφαρμόζεται και στον τομέα των κρασιών. Πιο συγκεκριμένα, η Επιτροπή υιοθέτησε έναν ξεκάθαρο κανονισμό ο οποίος σέβεται την αρχή της επικουρικότητας και μειώνει την περίοδο εφαρμογής. Αυτό θα επιστρέψει στην Επιτροπή να εστιάσει στα βασικά στοιχεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο χωρίς να ε, επαναλαμβάνει τους ίδιους ελέγχους που έχουν ήδη διενεργηθεί. Κάτι το οποίο θα είναι μια σαφής βελτίωση του συστήματος αλλά και της προστασίας των ενδιαφερόντων των παραγωγών. θα χρησιμεύσει και ως βάση για την κοινή αγροτική πολιτική 2020 για επιπλέον απλουστεύσεις στα πλαίσια ευθυγράμμισης των κανονισμών. Θα πρέπει να δράξουμε την ευκαιρία και ελπίζει η Επιτροπή το Κοινοβούλιο να α, ενστερνιστεί πλήρως την κατεξουσιοδότηση αυτήν πράξη. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Ανόφιλε για την παρουσίαση. Ο κύριος Δικάστρο έχει το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ και θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την DG Agri, ιδιαίτερως τον ε, Διευθυντή Όφρο, για τις εξηγήσει του όσο αφορά εμένα προσωπικά. Το διορθωτικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διευκρινίζει απολύτως ε, και τις δικές μας ανησυχίες, τα δικά μας μελήματα και έτσι αποσύρω εγώ τουλάχιστον την αντίρρηση και υποστηρίζω το ταχύτερο δυνατό να περάσουμε, την ιδέα από ταχύτερο δυνατό να περάσουμε στην κατεξοδότηση πράξη. Ευχαριστούμε κύριε Δεκάστρο. Ο κύριος Νταντά. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Είχα συζητήσει με τον ε, Παόλο πριν να γίνει αυτή η κίνηση. Είχα την ευκαιρία να συνομιλήσω και με τους εκπροσώπους της αρμόδιας ε, Γενικής Διεύθυνσης και θέλω να τους ευχαριστήσω που αφουγκράστηκαν τα κοινοβούλιο εγκαίρως ε, και με ικανοποιητικό τρόπο και έτσι δεν χρειάζεται να κάνουμε τσάπα δουλειά. Ευχαριστώ. Όντως, κύριε Νταντά, η σωστή συνεννόηση καταλήγει και σε καλές λύσεις. Ο κύριος Δόρφμαν. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρόκειται για μια κατεξουδότηση πράξη που έχει πολύ μεγάλη σημασία για τον ε, αμπελοϊνικό τομέα. Όπως είπαν και οι συνάδελφοι, μπορέσαμε να διευκρινίσουμε ζητήματα που είχαν ε, μείνει εκρεμή ε, αυτές τις τελευταίες εβδομάδες. Λοιπόν, τα επιλύσαμε και νομίζω ότι όπως είπε και ο κύριος Φωνόφερ μπορούμε πλέον με το νέο έτος να δούμε τους νέους κανόνες κυρίως για τη διαδικασία της αναγνώρισης της προστατευόμενης γεωγραφικής προέλευσης που είναι πολύ σημαντική. Έχουμε δει μια κάποια βραδύτητα και περιπλοκότητα στις διαδικασίες εδώ στις Βρυξέλλες για τα θέματα αυτό. Γι' αυτό είναι καλό το ταχύτερο δυνατό να επιστρέψει η δυνατότητα της ε, ρύθμισης με τις ε, κατεξοδότητες συμπράξεις ε, στα κράτη για να προχωρούμε ταχύτερα. Πρόκειται άλλωστε και για την πεμπτουσία των κατεξοδότης συμπράξεων, για να μην χρειάζεται να ταλαιπωρείται και να χάνει χρόνο ο παραγωγός. Άρα το, καλύτερο, το ταχύτερο δυνατό είναι και το καλύτερο. Ευχαριστούμε κύριε Ντόρφμαν. Δεν ξέρω αν ο ε, κύριο Ονόφρε, εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θέλει να δευτερολογήσει. Όχι από ό,τι βλέπω. Σα ευχαριστώ. Όντω είχαμε καταπληκτική συνεννόηση. Αυτό είναι ο σωστό δρόμο. Παίρναμε στο επόμενο σημείο, μια και διεκπαιρεώσαμε το 5. Προχωράμε στο 6. Περιμένουμε το εκπρόσωπο του ελεκτικού συνεδρίου, τον κύριο Βοητσεχόφσκι που είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου. Περιμένουμε να έρθει ο κύριος Βοητσεχόφσκι. Θα μας παρουσιάσει την ειδική έκθεση παριθμών 31 κάθετος 2018 με τίτλο «Καλή διαβίωση των ζώων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ φιλόδοξων στόχων και υλοποίησης στην πράξη». Quiero dar en la bienvenida en nombre. Θα ήθελα λοιπόν εκ μέρου τη ε, Επιτροπή Γεωργία και Ανάπτυξη Πέθρου να καλωσορίσω τον πρώην συνάδελφό μα τη Επιτροπή Άγκρη και νυν μέλο του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου, τον αγαπητό φίλο και πρώην αντιπρόεδρο τη Επιτροπή Άγκρη, Γιάννου Βοητσεχόφσκι ανέλαβε την εκπόνηση της ειδική έκθεσης του Ελεκτικού Συνεδρίου, μιας έκθεσης που ενδιαφέρει ιδιαίτερο στην Επιτροπή μας, μια και αφορά την, την ευζοία, την καλή μεταχείριση, την καλή διαβίωση των ζώων. Και μάλιστα ε, έχουμε και μια εφαρμοστική έκθεση που ετοιμάζει η Επιτροπή με συμμετοχή των ε, Επιτροπών Περιβάλλοντος και Μεταφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με βάση τον κανονισμό του 2005 της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κύριος Ντόρφμαν είναι ο εισηγητής μας για την έκθεση αυτή. Και μάλιστα η ειδική έκθεση φαίνεται ότι είναι πιο ευρία, έχει μεγαλύτερη εμβέλεια, δεν καλύπτει μόνο τη μεταφορά των ζώων, αλλά και την διαβίωση στις κτηνοτροφικές μονάδες και τη σφαγή. Μάλιστα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει από τις υψηλότερε προδιαγραφές και πρότυπα για την ευζοία στον κόσμο. Και μάλιστα είναι τμήμα της κοινή γεωρικής πολιτικής, ε, συμβάλλοντας στο στόχο της καλή μεταχείρισης των ζώων, χάρη στην πολλαπλή συμμόρφωση. Και επίσης χρηματοδοτεί δραστηριότητες και προγράμματα για την καλή μεταχείριση των ζώων στις ε, αναπτυσσόμενε αγροτικέ περιοχέ. Στο παρελθόν όμω είχαμε κάποια προβλήματα με την εφαρμογή των σχετικών προτύπων και προδιαγραφών τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την καλή μεταχείριση των ζώων. Αυτό είναι το θέμα που θα μα απασχολήσει σήμερα κατά την εξέταση τη ειδική έκθεση του Ελεκτικού Συνεδρίου. Η ειδική αυτή έκθεση εξετάζει το θέμα της καλής διαβίωσης των ζώων στις κτηνοτροφικές μονάδες και την γενική εφαρμογή της τελευταίας στρατηγικής για την ευζοία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2012-2015 και επικεντρώνεται στους δύο πρωταρχικούς στόχους, την υλοποίηση ελάχιστων προδιαγραφών και την βελτιστοποίηση των συνεργειών με την κοινή γεωργική πολιτική. Θα δώσω τώρα αμέσω ε, το λόγο στον κύριο Βοτσεχόφσκι. Δεν ξέρω αν προφέρω σωστά το όνομά και συγγνώμη αν κάνω λάθος, για να μας εξηγήσει λεπτομεριακά τα πορίσματα της ειδικής αυτής έκθεσης και θα ακολουθήσει συζήτηση. Ελπίζω να έχουμε ενδιαφέρουσα συζήτηση και ζωηρή συζήτηση για το θέμα αυτό τη ευζοία, γιατί είναι από τα πιο προσφυλή στην Επιτροπή μα. Γι' αυτό και θα δώσω το λόγο στον κύριο Βοητσεχόφσκι για ένα τέταρτο. Thank you, Madam President. Ευχαριστώ, κύρια Πρόεδρε, αγαπητά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι τιμή μου να σας παρουσιάζω σήμερα τα πορίσματα του ελέγχου του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για την καλή διαβίωση των ζώων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι η πρώτη φορά που οι ελεγκτές Ευρωπαϊκής Ένωσης εστιάζουν απολύτως στην καλή μεταχείριση των ζώων. Ο Μαχάτ Μαγκάντι ε, εξέφρασε μια σκέψη κάποτε ότι το μεγαλείο ενός έθνους και η ηθική του πρόοδος μπορεί να φανεί από τον τρόπο που φέρονται στα ζώα. Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το γνωρίζουν αυτό και όλο και περισσότερο ενδιαφέρονται για την καλή μεταχείριση και την ευζοία των ζώων. Το σκεπτικό της καλής κατάστασης των ζώων είναι εγγεγραμμένο στο άρθρο 13 της Συνθήκης Λειτουργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης που αναγνωρίζει τα ζώα ως νοήμωνα όντα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάποια από τα υψηλότερα στάνταρ σε ό,τι αφορά την ευζοία των ε, ζώων, όπως είπε και προηγουμένως η Πρόεδρος, που περιλαμβάνουν και προδιαγραφές για την ε, μεταφορά και τη σφαγή. Ο έλεγχος αυτός εστιάζει στα ζώα σε φάρμες. Επομένως, πολύ συχνά αναφέρεται στην νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξετάζουμε τα ζώα κτηνοτροφίας λόγω του κινδύνου του ότι μπορεί να μην τα μεταχειρίζονται σωστά, γιατί η καλή κατάσταση των ζώων πολλές φορές δεν συνάδει με τα οικονομικά συμφέροντα. Καθώς επίσης και η διάρκεια της ζωής των ζώων στη φάρμα, ο έλεγχος επίσης καλύπτει τη μεταφορά και τη σφαγή εξετάσαμε τη γενική εφαρμογή της στρατηγικής καλής, διαχείρισης των, καλής μεταχείρισης των ζώων, εστιάζοντας σε δύο στόχους. Πρώτα απ' όλα τη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές και τις συνεργίες με την κοινή αγροτική πολιτική. Εξετάσαμε α, σε πέντε κράτη-μέλη την καλή μεταχείριση των ζώων. Στη Γερμανία, στην Γαλλία, στην Ιταλία, την Πολωνία και τη Ρουμανία. Ο έλεγχο μα έδειξε ότι η Επιτροπή και τα κράτη-μέλη έχουν επιτύχει να ασχοληθούν, να εστιάσουν σε κάποια από τα ζητήματα καλής μεταχείρισης των ζώων μέσω ενός συνδυασμού κατευθυντήριων γραμμών και α, με τον επιβάλλουν κάποιες δράσεις. Α, τα σημεία α, επιτυχίας έχουν να κάνουν με τους κλοβούς για όρνηθες. Η Επιτροπή πολλές φορές καθυστέρησε να ασχοληθεί με τα προβληματικά σημεία. Σε πολλές περιπτώσεις ε, διαπιστώσαμε αδυναμίες ό,τι αφορά την εφαρμογή των ελάχιστων απαιτήσεων, ε, οι οποίε σε πολλέ περιπτώσει καθυστέρησαν να εγγραφούν στην νομοθεσία μέχρι και 18 χρόνια. Δυστυχώ οι αδυναμίε παραμένουν σε κάποιε περιοχέ, κυρίω σε ό,τι αφορά τα χειροστάσια, την έλλειψη συμμόρφωση με του κανόνε για την μακρά μεταφορά και την χρήση των διαδικασιών σφαγής. Πιο συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά τους κανόνες αναισθητοποίησης για την ε, σφαγή. Πιο συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά την, την αναισθητοποίηση για την σφαγή, δεν υπάρχουν γενικές γραμμές σε ό,τι αφορά την σφαγή. Αυτό που διαπιστώσαμε είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν αρκετές παρακαμπτηρίες οδοί. Για παράδειγμα, στη Γερμανία υπήρχε μια ειδική διαδικασία για να δικαιολογήσει την διαδικασία ασφαγής. Ακόμα και οι πιο υψηλές προδιαγραφές μεταχείρισης των ζώων δεν θα αλλάξουν την κατάσταση αν τα συστάματα ελέγχου δεν είναι αποτελεσματικά. Διαπιστώσαμε βέλτιστες πρακτικές, κυρίως σε ό,τι αφορά τη συνέπεια με τους επίσημους ελέγχους ή την ε, πρόληψη σύγκρουση συμφερόντων. Παρ' όλα αυτά, διαπιστώσαμε και αδυναμίες στα συστήματα ελέγχου των κρατών μελών πιο συγκεκριμένα αφορούσαν α, στους συγκεκριμένους ελέγχους, κυρίως στον τομέα μεταφοράς ζωντανών ζώων. Για παράδειγμα, ο έλεγχος των οδών στην Πολωνία, που δεν υπήρχε πρόσβαση στο σύστημα Traces. πολλές φάρμες εξαιρούνται από τους επίσημους ελέγχους, παρόλο που αντιπροσωπεύουν ένα μεγάλο κομμάτι της κτηνοτροφίας, πιο συγκεκριμένα στην Ιταλία και στην Ρουμανία, η χρήση πληροφοριών από καταγγελίες σε ορισμένα κράτη-μέλη. Διαπιστώσαμε ότι μόνο δύο από τα κράτη-μέλη που επισκεφτήκαμε, η Πολωνία και η Ρουμανία, έχουν διαδικασίες που έχουν να κάνουν με την καταγγελία παραπώνων. Κανένα από τα κράτη-μέλη δεν εφαρμόζει ένα κεντρικό κατάλογο βάση δεδομένων που να δίνει μια γενική εικόνα των βασικών τομέων ανησυχία σε ό,τι αφορά την καλή μεταχείριση των ζώων. Η στρατηγική καλή μεταχείριση των ζώων τη Επιτροπή 2012-2015 αναγνώρισε την ανάγκη βελτίωση συνεργειών μεταξύ τη καλή μεταχείριση των ζώων και των εργαλείων τη ε, κοινή αγροτική πολιτική κυρίως μέσω της α, α, γεωργικής ανάπτυξης. Ο μηχανισμός α, συμμόρφωσης θα επιτρέψει στους κτηνοτρόφους να μπορέσουν να επιτύχουν υψηλότερες προδιαγραφές. Ένα από τα βασικά σημεία της έκθεσής μας είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει καλύτερη σύνδεση μεταξύ των διαφόρων τομέων εφαρμογής της πολιτικής. Τα κράτη-μέλη έχουν γενικά θέσει αρκετούς κανόνες σε ό,τι αφορά τους ελέγχους για την καλή μεταχείριση των ζώων. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει περιθώριο βελτίωσης των επίσημων ελέγχων. Υπάρχουν επίσης α, αρκετές περιπτώσεις όπου έχουν επιβληθεί α, πρόστιμα τα οποία δεν ήταν αναλογικά με τις α, παρατυπίες που διαπιστώθηκαν. Η αξιολόγησή μας είναι ότι η καλή μεταχείριση των ζώων θα μπορούσε να έχει εξαιρετικά αποτελέσματα πέρα από αυτά που προβλέπουν οι ελάχιστες απαιτήσεις. Παρ' όλα αυτά, τα μέτρα αυτά δεν, ιδίως ό,τι αφορούν τα μέτρα της αχυροστρομής. Παρόλα αυτά, τα μέτρα αυτά δεν χρησιμοποιήθηκαν ευρέως. Στην Γαλλία η επιλογή αυτή ήταν αντίθετη με την εθνική στρατηγική της καλής μεταχείρισης των ζώων, η οποία δεν επέτρεπε την ε, χρησιμοποίηση πόρων. Για να βελτιώσουμε την κατάσταση, κάναμε μια σειρά από συστάσεις. Πρώτα απ' όλα, αξιολόγηση της στρατηγικής καλής διαχείρισης των ζώων και εξέταση του πώς μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τα πορίσματα, για παράδειγμα σε ό,τι αφορά την νομοθεσία. Δεύτερον, ανάπτυξη μιας ε, στρατηγικής επιβολής, ώστε να μειώσουμε το χρόνο εφαρμογής των συστάσεων της Επιτροπής από τα κράτη-μέλη, ούτως ώστε τα προβλήματα που επιμένουν να μπορέσουν να εξαλειφθούν βελτίωση του συντονισμού ανάμεσα στους επίσημους ελέγχους και την πολλαπλή συμμόρφωση και τέλος χρήση της αγροτικής ανάπτυξης, ώστε να μπορέσουμε να επιτύχουμε καλύτερα τους στόχους μας ε, μέσω κυρίως της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και δίνοντας στους κτηνοτρόφους ε, περισσότερα κίνητρα, ώστε να μπορέσουν να βελτιώσουν την, ε, την μεταχείρισή τους απέναντι στα ζώα. Κυρίες και κύριοι, θέλω να υπογραμμίσω τα πιο σημαντικά ερωτήματα τα πιο σημαντικά ερωτήματα για σας είμαστε στην αρχή της συζήτησης που αφορά την κοινή αγροτική πολιτική. Και ένα ερώτημα που είναι πολύ σημαντικό έχει να κάνει με το ερώτημα 14 για το α, πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης. Και είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο το οποίο έχει να κάνει και με την βελτίωση από πρακτική άποψη της ευζοίας των ε, ζώων κτηνοτροφίας. Σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, την αχυρόστρωση για τα ή για παράδειγμα τους βαθμούς παστερίωσης τα θερινά βοσκοτόπια. Και εδώ πέρα μιλάμε για, την, για όχι κτηνοτροφία σε βιομηχανικό επίπεδο. Πρόκειται για ένα προϋπολογισμό 1,5 δισεκατομμυρίου. Ο πιο σημαντικός εταίρος ήταν η Ρουμανία, η οποία χρησιμοποίησε περίπου 30% της χρηματοδότησης αυτής. 18 κράτη-μέλη χρησιμοποίησαν το μέτρο αυτό. Είναι περισσότερα από ό,τι προηγουμένως, περισσότερα από το πρόγραμμα 2007-2008. Ήταν 15 κράτη-μέλη που χρησιμοποίησαν το μέτρο αυτό προηγουμένως. Είναι ένα πολύ συγκεκριμένο εργαλείο το μέτρο αυτό για τη βελτίωση της καλής μεταχείρισης των ζώων. Ένα δεύτερο πρόβλημα είναι το σύστημα ελέγχου, το οποίο θα πρέπει να βελτιωθεί. Κυρίως ό,τι αφορά το συντονισμό των ελέγχων πολλαπλής συμμόρφωσης. Το πιο, ένα πολύ σημαντικό ζήτημα είναι η σφαγή χωρίς νάρκωση, χωρίς αναισθητοποίηση. Όταν ε, ήμουν κι εγώ μέλον, μέλος της Επιτροπής αυτής, ήμουν αντιπρόεδρος της Επιτροπής αυτής, ήμουν εισηγητής του κανονισμού που αφορά στην σφαγή, που συζητήθηκε το 2009 στη σφαγή των ζώων. Και αυτό που συζητήσαμε τότε είναι ότι η σφαγή χωρίς νάρκωση θα πρέπει να είναι η εξαίρεση μόνο σε ε, περιπτώσεις που επιβάλλεται από θρησκευτικές πρακτικές θα πρέπει να χρησιμοποιείται. Τώρα βεβαίω υπάρχουν διαφορετικές ε, πρακτικές στα κράτη-μέλη. Για παράδειγμα είναι πολύ αυστηρή στη Γερμανία, στην Πολωνία είναι πιο ευέλικτη. Στην Πολωνία είναι ειδική περίπτωση, γιατί ε, δύο χρόνια πριν υπήρχε απόλυτη απαγόρευση της σφαγής χωρίς νάρκωση, το συνταγματικό δικαστήριο αποφάσισε ότι η απαγόρευση αυτή ήταν ενάντια στην θρησκευτική ελευθερία. Το ερώτημα όμως αυτό για τη συζήτησή μας. Έχουμε τον ίδιο κανονισμό αλλά διαφορετικές πρακτικές στα κράτη-μέλη και πιστεύω ότι αυτό θα πρέπει να αλλάξει. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε Είναι μόνο η αρχή, αλλά είμαστε εδώ για να απαντήσουμε σε ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Βοητσεχόφσκι. Το λόγο έχει τώρα ο εισηγητής μας, ο εισηγητής στην έκθεση πρωτοβουλίας, ο κύριος Ντόρφμαν. Τζον Ντόρμαν. Ο Τζον Ντόρμαν, συγγνώμη. Γιατί έχετε το ίδιο επίθετο. <laughs> και έτσι δεν το, δεν το πρόφερα και καλά. Ντόρφμαν ο ένα, Ντόρμαν ο άλλο. Ντόρμαν του προφέρω και του δύο. Ο κύριο Τζον Ντόρμαν είναι ο εισηγητή πάντω. Ευχαριστώ πολύ. Εδώ μου λέτε να σας κάνω την παρουσίαση για το θέμα της μεταφοράς των ζώων των ζώων. Αυτό μου λέτε. Συγγνώμη, μπερδεύτηκα, μπερδεύτηκα πάλι. Θα σας δώσω το λόγο για να μας σχολιάσετε αν θέλετε την έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου. Μετά θα περάσουμε στη συζήτηση για τη δική σας έκθεση. Ε, εντάξει, ευχαριστώ λοιπόν. Και θα ήθελα να πω ότι χαίρομαι που διαπιστώνω από τα όσα άκουσα ότι δουλεύουμε στην διακατεύθυνση στο ίδιο επίπεδο για να βελτιώσουμε την ευημερία των ζώων και σημειώνω ότι είναι όνειδος ότι έχουν διαφορετικές επιλογές ακολουθήσει τα κράτη-μέλη. Θα κοιτάξουμε λοιπόν να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε από εδώ και μπρος. Μέσα από την έκθεση θα δώσουμε προτάσεις. Πάντως είναι πολύ θετικό το ότι από ό,τι μας λέτε μπορούν να γίνουν κάποια πράγματα. Μπορούμε δηλαδή κάποια από τα κονδύλια που ε, διατίθενται για τον τομέα αυτό να στοχεύσουν στη βελτίωση της ευημερίας των ζώων για το μέλλον. Προσβλέπω λοιπόν σε μια επικοδομητική συζήτηση για το τι συγκεκριμένα μπορούμε να κάνουμε. Και συγκεκριμένα όταν μιλούμε για γεωργικές ενισχύσεις, μήπως πρέπει να τις στοχεύσουμε στην Ευημέρεια των ζώων. Χαίρομαι που και το ελεγκτικό συνέδριο αντιμετωπίζει με πολύ μεγάλη σοβαρότητα το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Ντόρμαν. Και πάλι για την έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου, το λόγο κυρία Σράιερ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Με μεγάλο θαυμασμό παρακολούθησα την παρουσίαση και ξεπλάγιν γιατί με όλη την προσοχή που αφιέρωσα στην ομιλία του κυρίου από το Ελεκτικό Συνέδριο δεν άκουσα να αναφέρει καθόλου τις κάτω Είναι όλα ρόδινα εκεί ή συμβαίνει κάτι άλλο, γιατί την γνωρίζω την κατάσταση αρκετά καλά στις κατοχώρες. Βεβαίως υπάρχει υποχρέωση για την αναισθητοποίηση πριν από τη σφαγή. Πιστεύουμε ότι έπρεπε να είναι αυτονόητο να συμβαίνει πάντοτε. Και για τις εξελίξεις για το μέτρο υπαριθμών 14, η ερώτησή μου θα είναι πώς μπορούμε να ε, το αναπτύξουμε περαιτέρω. Έχουμε καταθέσει τροπολογίες, είχαμε προθεσμίω στις 3, ωστόσο η κατάσταση που επικρατεί στην κάθε χώρα διαφέρει από αυτήν μιας άλλης χώρας για την ε, αχυροστρομνή για χείρους. Υπάρχουν ε, ε, γεωργικές εκμεταλλεύσεις που ακολουθούν το σύστημα αυτό της χειροστρομής. Αλλά όμως έχουν υποδαπέδια θέρμανση. Και αυτό μπορεί να αποδεικνύεται καταλληλότερο για τους χείρους. Στο Λάρνγκεν που ήμουν την προηγούμενη εβδομάδα μου κάνανε μια παρουσίαση και μου εξήγησαν ότι η στάβληση των αγελάδων δεν είναι πάντα ε, κάτι το αρνητικό για τα ζώα. Δεν σημαίνει ότι τους κάνει πάντα κακό. Έτσι λοιπόν προτείνεται ως σύσταση, ως ε, προτιμόμενη ε, μεταχείριση, αλλά πρέπει να δούμε και τις ιδιαίτερες ε, περιστάσεις και από ευρωπαϊκής πλευράς πρέπει να μην μιλούμε μόνο για, σε όρους οικονομικού ή τιμών για το γεωργό. Γιατί αν ακολουθήσουμε αυτή τη λογική κατά τρόπο ομοιόμορφο όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα έχουμε καταστρέψει τον ανταγωνισμό. Ευχαριστούμε κυρία Σράιερ. Θα ήθελα να περιορίσω το χρόνο ομιλία στο δίλεπτο. Ο κύριος Χόισλινγκ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πουσκόφσκι για την έκθεση. Ε, ξεκάθαρα αυτό που μας είπατε. Πρώτη ερώτηση, διαφορετικές προδιαγραφές στην Ευρώπη. Υπάρχουν κράτη τα οποία αξιοποιούν την ε, παρέκκληση ε, όπως ε, η Γερμανία και για την κοπή της και για την για τον ευνοχισμό χωρίς ε, αναισθητοποίηση. Βλέπουμε ότι αυτό γενικεύεται. Βλέπουμε ότι υπάρχουν διατάξεις οποίες τα κράτη ερμηνεύουν κατά διαφορετικό τρόπο. Πώς λοιπόν μπορούμε να τα ρυθμίσουμε όλα αυτά και πόσο ακόμα μπορούμε να ερχόμαστε στην ίδια κατάσταση. Επίσης, είπατε ότι υπήρξαν κράτη τα οποία δεν αξιοποιούν την δυνατότητα χρηματοδότησης της ε, ευημερίας των ζώων από το δεύτερο πυλώνα. είναι ξεκάθαρο ότι σε πολλούς τομείς ε, έχουν περιθώριο βελτίωσης, για να μην πω μεγάλο περιθώριο βελτίωσης προδιαγραφές. Έτσι λοιπόν δεν νομίζω ότι μπορούμε να περιοριστούμε μόνο σε μια εκούσια συμμόρφωση. Πρέπει να αλλάξουμε κάτι και στα σοβαρά. Τρίτη ερώτηση, έλεγχη. Είπατε ότι υπάρχουν διαφορετικές και, και ε, επιθεωρήσεις. Είπατε ότι υπάρχουν διαφορετικές προδιαγραφές στην Ευρώπη για το τι είναι επιθεώρηση και πώς διεξάγεται. Φερρυπίν. Εάν γίνεται επιθεώρηση σε μια ε, γεωργική εκμετάλλευση στη Βαβαρία μια φορά στα 20 χρόνια, πώς θα πρέπει να το κοιτάξουμε πιο προσεκτικά. Και στην σφαγή πάλι. Να και το αναφέρατε. Ε, είχα στο μυαλό μου βέβαια και την τελετουργική σφαγή για θρησκευτικού λόγους, αλλά ξέρουμε ότι έχουν κλείσει ε, κάποια σφαγεία και μάλιστα όχι μόνο προσωρινά στη Γερμανία, γιατί τακτικά διαπιστωνόταν ότι όχι μόνο γινόταν σφαγιζόν χωρί χωρίς την αισθητοποίηση, αλλά και σφαγιζόν που δεν έπρεπε να έχουν σφαγή. Άρα υπήρχαν σοβαρές παραβιάσεις της ε, νομοθεσίας. Είχαμε και μια ε, ταινία από βίντεο που προέκυψε και έδωσε στοιχεία. Θα ήθελα λοιπόν σε αυτές τις διαδικασίες τι μπορείτε να δείτε σαν δυνατότητες βελτίωσης. Ευχαριστούμε κύριε Χόισλινγκ. Σας υπενθυμίζω το δίλεπτο που έχετε στη διάθεση. Κυρία Νόιχλου. Ναι, ευχαριστώ πρόεδρε. Με συγχωρείτε που σηκώσα το χέρι. Την επόμενη έκθεση ήθελα εγώ. Ε, ευχαριστώ πολύ το ελεκτικό συνέδριο για την έκθεση. Καράτε τη διασύνδεση της ε, γεωργικής πολιτικής με τις άμεσες ενισχύσεις και τις ευημερίες των ζώων. Ε, τρία είναι τα κύρια θέματα που βλέπω να προκύπτουν από την έκθεσή σας. Η θέση των ζώων και η ευημερία τους μέσα στις εκμεταλλεύσεις. Θεωρείτε ότι η διαδικασία εκμετάλλευσης και κτηνοτροφίας στις Βρυξέλλα, στην Ευρώπη μπορεί να βελτιωθεί και αυτό από τους κτηνοτρόφους μπορούμε να το ζητήσουμε γιατί βλέπουμε μερικές φορές ότι υπάρχουν κτηνοτρόφοι οι οποίοι δεν έχουν καν κατάρτιση τέτοια. Ε, επίσης το θέμα της μεταφοράς των ζώων οι μεταφορικές επιχειρήσεις δεν θα έπρεπε περισσότερο να κληθούν να τηρήσουν τις προδιαγραφές, να υποχρεωθούν, γιατί υπάρχουν προδιαγραφές που όμως δεν ελέγχεται, όπως άλλωστε και εσείς ο ίδιος είπατε, δεν γίνονται επαρκείς ε, επιθεωρήσεις στον, στις μεταφορές των ζών. των ζώων. Για δε τη σφαγή υπάρχουν συνθήκες εργασίας για τους εργαζομένους εκεί, τέτοιες που να επιτρέπουν μία σφαγή με τον κατάλληλο τρόπο και βέβαια και την ανιστοποίηση. Όλα αυτά βλέπω εγώ από τα όσα μας είπατε και ε, συνοπτικά διαπιστώνω ότι μας λέτε πως έχουν τελείως διαφορετική θεώρηση και ερμηνεία τα κράτη-μέλη και εφαρμογή για τα αισθήματα της ευημερίας των ζώων. Πώς νομίζετε ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε νέες προδιαγραφές, πώς μπορούμε να αποφύγουμε την περαιτέρω στρέβλωση του ανταγωνισμού που προκύπτει από τη διαφορετική εφαρμογή ε, προδιαγραφών από τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κυρία eh, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς τον κύριο Βοητσεχόφσκι για την παρουσίαση της έκθεσης του Ενακτικού Συνεδρίου. Είναι η πρώτη φορά που το Ευρωπαϊκό, το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο ενέκυψε σε αυτό το θέμα της καλής μεταχείρισης των ζώων και η πρώτη έκθεση με το θέμα αυτό. Χαίρομαι για αυτή τη στροφή στα ενδιαφέροντα του Ελεκτικού Συνεδρίου. Ε, κανόνες έχουμε, αλλά δυστυχώς δεν εφαρμόζονται κατάλληλα. Και πραγματικά είναι συγκλονιστικό ότι τόσες πολλές χώρες δείχνουν τέτοια αδιαφορία για την καλή μεταχείριση των ζώων, παρά τις αυστηρές προδιαγραφές και τα πρότυπα που έχουμε. Έχουμε από τις αυστηρότερες προδιαγραφές και πρότυπα στον κόσμο για την καλή διαβίωση των ζώων, αλλά δυστυχώς δεν τα εφαρμόζουμε παντού. Αναφέρθηκε η απαγόρευση ακατάλληλων κλοβών για τις οτόκες όρνηθες. Ε, ε, οι αποφάσεις, οι αυτές έχουν ληφθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αλλά δεν εφαρμόζονται. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε από την αρχή της θητείας της ότι δεν είχε καμία πρόθεση να προτείνει νέα νέα νομοθετικά μέτρα για το εγγύς μέλλον. Έχω να σας υποβάλω μια ερώτηση. Πιστεύετε ότι θα συνεχίσουμε στην Ευρώπη να είμαστε πρωτοπόροι στα θέματα αυτά, γιατί βλέπω ότι χώρες όπως η Κίνα δεν μας μιμούνται, αλλά έχουν τις δικές τους διατάξεις και πρότυπα για την καλή διαβίωση των ζώων. Δεν είμαστε πια σκαπανεί πρωτοπόροι που ήμασταν στο παρελθόν. Οπότε θα είναι δύσκολο να εφαρμόσουμε και τη δική μας στρατηγική, γιατί φαίνεται ότι στερείται συγκεκριμένων στόχων. Έχει νόημα, κατά τη γνώμη σας, να αξιολογήσουμε την παλιά μας στρατηγική, αν δεν υπάρχει κανένα σχέδιο για νέα στρατηγική για τα θέματα αυτά. Σε αντίθεση με τα αιτήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ήταν υπέρ μιας νέας στρατηγικής. Υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των χωρών μελών και θα πρέπει να γεφυρώσουμε το κενό μεταξύ μιας φιλόδοξης νομοθεσίας και της πενιχρής ε, εφαρμογής της. Επίσης θέλουμε και οι νέες νομοθεσίες να είναι φιλόδοξες και αν δεν έχουν επιβληθεί κυρώσει ε, για τις τη ατασταλή, αυτό θα διορθωθεί. Να επιβληθούν κυρώσει και πρόστιμα. Είναι κρίμα να δρανεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ελπίζω να γίνει καλύτερος έλεγχος. Ο κύριο Κούσμιουκ, ευχαριστώ και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Βοητσεχόφσκι για την έκθεση του Ελεκτικού Συνεδρίου. Και από ό,τι κατάλαβα, ελέγχθηκε η κατάσταση της καλής μεταχείρισης σε τρεις παλιές χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε δύο από τις νέες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φυσικά υπάρχει διαφορά μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης παλιών και νέων σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των πολιτικών, γιατί οι νέε χώρε εφαρμόζουν τη νέα πολιτική από το 2014, ενώ οι παλιές χώρες μέλη υποφελήθηκαν από την κάπεδο και πάρα πολλά χρόνια. Στη σύγκριση μεταξύ των δύο κατηγοριών χωρών, πώς έχει η καλή μεταχείριση των ζώων. Πού είναι η καλύτερη κατάσταση ό,τι αφορά την καλή διαβίωση των ζώων, στις παλιές χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στις νέες, ή μήπως υπάρχει μια ισορροπία. Σε ό,τι αφορά τους μηχανισμούς που εφαρμόζουν παλιες χωρες μελη της ευρωπαικης ενωσης στις νεες η μηπως υπαρχει χώρες και τις α, ε, πενιχρές δαπάνες ε, του πρώτου πυλώνα. Είπατε για μία αιτία προβλέπετε 1,5 δισεκατομμύριο προπολογισμό για τα θέματα αυτά. Ελάχιστο, πενιχρό ο προπολογισμό. Γιατί είναι μικρό το ενδιαφέρον των κρατών μέλων ε, να εφαρμόσουν τέτοια προγράμματα και να τα, συμπεριλαμβάνουν, να τα συμπεριλάβουν στι εθνικέ πολιτικέ. Ή οφείλεται αυτό ο μικρό προπολογισμό στην αυστηρή προσέγγιση Ευρωπαϊκή Επιτροπή που δεν κρίνει επιλέξιμα αρκετά προγράμματα, εξού και μικρό αριθμό των προγραμμάτων που αποφελούνται από αυτά τα κονδύλια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Κουσμιούκ. Δεν ξέρω αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκπρόσωπο για τα θέματα αυτά και θέλει να λάβει το λόγο. Δεν βλέπω κανέναν, οπότε να δώσω το λόγο και πάλι στον καλεσμένο μας για να απαντήσει στις ερωτήσεις και να ολοκληρώσουμε αυτό το θέμα. Κύριε Βοτσιχόφσκι, έχετε και πάλι το λόγο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Mm. Θα απαντήσω στη μητρική μου γλώσσα που είναι τα πολωνικά. Ε, να απαντήσω στις ερωτήσεις της κυρίας Σράιερ καταρχήν για την Ολλανδία. Διαλέξαμε πέντε χώρες για να πραγματοποιήσουμε ελέγχους. Τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, τη Ρουμανία και την Πολωνία. Τρεις παλιές και δύο καινούριε. Εκεί έχουμε την πιο εκτεταμένη κτηνοτροφία. Αυτές οι πέντε χώρες έχουν περισσότερες, ε, περισσότερα ζώα εκτροφής από ό,τι οι υπόλοιπε. Αυτό ήταν το κριτήριο της επιλογής μας και οι κάτω χώρες δεν ήταν σε αυτή την κατηγορία. Φυσικά, κάναμε έλεγχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δεν κάναμε ειδικό έλεγχο των κάτω χωρών. Ελέγξαμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις δράσεις της όλα τα κράτη-μέλη, αλλά σε ό,τι αφορά τις συγκεκριμένους ελέγχους αφορούσαν τις πέντε χώρες μόνο. Σε ό,τι αφορά τη σφαγή, δεν μιλήσαμε για την τελετουργική σφαγή, μιλήσαμε μόνο για σφαγή χωρίς προηγούμενη αναισθητοποίηση. Γνωρίζουμε περί πρόκειται. Και φυσικά εδώ υπάρχουν και άλλα ζητήματα έχουμε προβλήματα γιατί είναι πολύ διαφορετικές οι πρακτικές και οι μέθοδοι της φαγής και δεν υπάρχει συγκεκριμένος ορισμός. Υπάρχει κάποια διάταξη, ή κάποια αρχή μάλλον, που καλό θα είναι να το τη λάβουν υπόψη τα κράτη-μέλη, αλλά δεν ε, είναι σαφές ποιες είναι οι θρησκευτικέ προϋποθέσεις. Δεν προσδιορίζεται κάτι τέτοιο αν υπάρχουν τέτοιες θρησκευτικέ απαιτήσει. και αν αυτές οι τελετουργικές σφαγέ εξυπηρετούν κάποιες τοπικές θρησκευτικές κοινότητες ή αφορούν και ζώα που θα εξαχθούν προς χώρες που επίσης απαιτούν τέτοιου είδους τελετουργική σφαγή. Οπότε πληρούνται οι υποθέσει για την εφαρμογή τη εξαίρεση ή όχι. Δεν είναι σαφέ αυτό από την κοινοτική νομοθεσία. Θα πρέπει λοιπόν να διευκρινιστούν αυτέ οι διατάξει, γιατί υπάρχουν πολλέ διαφορετικέ πρακτικέ. Και αφήνουμε τα ανθρωπιστικά στοιχεία. Μερικές φορές παραβιάζονται οι όροι του ισότιμου ανταγωνισμού, του θεμητού ανταγωνισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αφήνουμε του ανθρωπιστικού λόγου. Υπάρχουν μεγάλε διαφορέ πρακτικέ που χρησιμοποιούν τα κράτη-μέλη. Και αυτό είναι ένα από τα θέματα που χρήζουν περαιτέρω συζήτηση, ανάλυση και ίσω και κάποια νομοθετική μεταρρύθμιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το ανέφερε και ο κύριος Χόισλινγκ αυτό το σημείο. Εξού και η δική μου απάντηση. Όλα αυτά τα θέματα της φαγή και κυρίως της λειτουργικής σφαγής χρήζουν πολύ πιο διεξοδική συζήτηση. Και υπό ποιες προϋποθέσεις επιτρέπουμε τέτοια σφαγή χωρίς αρεστητοποίηση. Στη Γερμανία ελέξαμε στη Ρινανία Βεσφαλία κάποιε κάποιες κτηνοτροφικές μονάδες αλλά αναλύσαμε τη γερμανική νομοθεσία γενικώ που είναι πολύ περιοριστική και είναι ελάχιστε οι σφαγέ που γίνονται χωρί αναισθητοποίηση στη Γερμανία. Αντίθετα, στην Πολωνία Σχεδόν είναι άγνωστη αυτή η πρακτική της αναισθητοποίησης ε, και δεν γνωρίζουμε πόσες, ε, πόσα σφαγεία εφαρμόζουν τέτοιες ε, μεθόδους. Αν γίνεται σφαγή με ή χωρίς νάρκωση. Δεν έχουμε στοιχεία για την Πολωνία. Πολλά. Ή δεν ξέρουμε αν κάποιες σφαγές γίνονται με βάση κάποιες τελετουργικές απαιτήσεις ή μερικές φορές και ε, για κάποια άλλα κριτήρια. Όλα αυτά χρήζουν ε, διεξοδική συζήτηση και κάποιες νομοθετικής αναθεώρησης, γιατί είναι κάπως αόριστα και ε, συγκεχημένα τα θέματα. Αυτά και επισημαίνουμε τα κενά που υπάρχουν εδώ στην νομοθεσία ως προς τους αφισορισμούς. Ευχαριστώ και την κυρία Χάζεκαμπ για τις παρατηρήσεις που μας έκανε και την θετική υποδοχή που επιφύλαξε στην έκθεση του Διαλεκτικού Συνεδρίου. Υπάρχει όμως πρόβλημα, όπως είπαμε, με την εκτέλεση, την εφαρμογή των κοινοτικών διατάξεων για την καλή μεταχείριση των ζώων. Οπότε θα πρέπει να γίνουν προσπάθειες όχι για την ε, θέσπιση νέων νομοθετικών διατάξεων, αλλά για την βελτίωση του συστήματος ελέγχου, ώστε να υπάρχει πιο αποτελεσματικό σύστημα ελέγχου για να εξακριβωθεί η τήρηση των υψηλών προδιαγραφών και προτύπων που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την καλή μεταχείριση των ζώων. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να είναι πρωτοπόρο σε θέματα καλής μεταχείρισης των ζώων, εξακολουθεί να παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο. Θεωρούμε ότι είμαστε ακόμη πρωτοπόροι και πολλές χώρες προσπαθούν να μας φτάσουν και χαιρόμαστε γι' αυτό. Θέλουμε να δώσουμε το καλό παράδειγμα και να ευαισθητοποιήσουμε σε παγκόσμια κλίμακα τις χώρες για την καλή μεταχείριση των ζώων, αλλά οι καλές προδιαγραφές και αυστηρές προδιαγραφές ε, δεν ε, διαδραματίζουν το ρόλο τους αν δεν εφαρμόζονται στην πράξη. Ο κύριος Κουσμίουκ με ρώτησε για τη διαφορά παλιών και νέων χωρών. Πέντε χώρες ελέγξαμε, δύσκολο να κάνουμε ε, κάποια ιεράρχηση και στις πέντε χώρες είχαμε και καλές και λιγότερο καλές πρακτικές. Δεν υπάρχουν ιδιαίτερες διαφορές στις επιδόσεις. Πάντως, σχετικά αρκετές καλές πρακτικές βρήκαμε στην Ιταλία. Στην Ιταλία γενικώ και στη Σαρδινία ειδικώ είχαμε πολύ θετικές εμπειρίες και πολύ καλές πρακτικές ε, για την εφαρμογή του μέτρου 14, 14 Επίση, αναλύσαμε το θέμα τη σύγκρουση συμφερόντων, δηλαδή η κτηνιατρική έλεγχη είναι απαλλαγμένη από τη σύγκρουση συμφερόντων. Στην περίπτωση αυτή, στην Ιταλία είχαμε πολύ θετικέ λύσει ε, αποκλείοντα τη σύγκρουση συμφερόντων. Στην Ιταλία όμω είχαμε άλλο πρόβλημα. 13 χρόνια χρειάστηκαν για να μεταφερθεί στην εσωτερική Ιταλική Ένωμη Τάξη η οδηγία τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την αποχρέωση, για την η υποχρέωση της ε, υποχρεωτικής, ε, του υποχρεωτικού ξεποπουλιάσματος των πουλερικών. 13 χρόνια χρειάστηκε να περάσουν για να εφαρμόσει η Ιταλία τη σχετική ε, νομοθεσία. Οπότε υπάρχουν κάποιες διαφορές, αλλά δεν κάναμε... Δεν καταρτήσαμε πίνακα βαθμολόγησης ποιος είναι ο καλύτερος μαθητής και ποιος ο χειρότερος από τις πέντε χώρες που ελέγξαμε. Πάντως, ό,τι αφορά την, το μέτρο υπαριθμών 14 και την εφαρμογή του, αυτό είναι εθνική επιλογή. Τα κράτη-μέλη έχουν τη διακριτική ευχέρεια να αποφασίσουν αν θα εφαρμόσουν αυτές τις δραστηριότητες του μέτρου 14. Μερικές χώρες τις εφάρμοσαν, άλλες όχι. Γενικώ πάντως υπήρχε κάποιος κίνδυνος διπλής χρηματοδότησης από το μέτρο 14 να εφαρμοστούν ε, μέτρα που χρηματοδοτήθηκαν και από ένα κονδύλιο για την ποιότητα των τροφίμων ή την ποιότητα των ζωοτροφών. Υπήρξαν κάποιοι τέτοιοι κίνδυνοι, πάντως πιστεύω ότι αυτό το μέτρο, το μέτρο 14 και σχετικές δράσεις ε, είναι η καλύτερη μέθοδος για να δώσουμε κίνητρα στους ακτινοτρόφους για να εφαρμόσουν ε, τις αυστηρές προδιαγραφές. Μερικές φορές και με πρόστιμα βέβαια και με κυρώσεις αλλά νομίζω ότι καλύτερα αποτελέσματα δίνουν τα κίνητρα για την ε, αναβάθμιση και την ε, καλύτερη εφαρμογή των προδιαγραφών. Γιατί μερικές φορές η καλή μεταχείριση των ζώων αποβαίνει και προς όφελος της καλής κατάστασης των κτηνοτρόφων. Είναι προ το συμφέρον και των κτηνοτρόφων η καλή διαβίωση των ζώων και σε καμία περίπτωση κάτι τέτοιο δεν μειώνει την ανταγωνιστικότητα των κτηνοτρόφων. Το αντίθετο, ε, βελτιώνεται η ανταγωνιστικότητα των κτηνοτρόφων χρησιμοποιώντας ε, κίνητρα για την ε, αναβάθμιση των προδιαγραφών της καλής μεταχείρισης. Και πρέπει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δίνει κίνητρα, αλλά τα κράτη-μέλη έχουν την ευχαίρεια επιλογής των συγκεκριμένων δράσεων για την υλοποίηση αυτών των κινήτρων προς τους κτηνοτρόφους. Και μία ακόμη ερώτηση. Πολύ ενδιαφέρουσα ήταν η ερώτηση της κυρίας Μίλλερ για, για τη μεταφορά και αν θα πρέπει να ενισχύσουμε τις απαιτήσει μας από τις μεταφορικές εταιρείες. Ίσως, ίσως ο κανονισμός που αφορά τις μεταφορές προσδιορίζει με σαφήνεια τους όρους και τις προϋποθέσεις της μεταφοράς των ζώων. Υπάρχει όμως άλλο πρόβλημα κατά τη γνώμη με τη μεταφορά γιατί και τι προκαλεί ε, μεταφορές σε τόσο μεγάλες αποστάσεις. Γιατί χρειάζονται να μεταφέρουμε ζώα σε τόσο μεγάλες αποστάσεις. Και χαίρομαι που ο κύριος Ντόρμαν στην, στην έκθεση του αναφέρει σε ένα από τα 15 σημεία την ανάγκη περιορισμού των τόσο μεγάλων αποστάσεων μεταφορών. Και να δούμε γιατί γίνονται τέτοιε μεταφορές σε τόσο μεγάλες αποστάσεις, ποιο πληρώνει το κόστος ε, τέτοιων μεταφορών. Συμφέρει να μεταφέρουμε ζώα σε τόσο μεγάλες αποστάσεις. Και μάλιστα ήμουν παρόν ε, στην ακρόαση που οργάνωσε ο κύριος Ντόρμαν για το θέμα αυτό και εκεί ακούσαμε πολύ ε, δραματικά αποτελέσματα για τη μεταφορά ζώων από την Ιρλανδία προς τη Μέση Ανατολή ολόκληρα κοπάδια που μεταφέρονταν από την Ιρλανδία στη Μέση Ανατολή. Συμφέρουν τέτοιε μεταφορέ σε τόσο μεγάλο κόστο. Ποιο αναλαμβάνει το κόστο τέτοιων μεταφορών, Γιατί πολλά λέμε για την ατμοσφαιρική ρήπανση και η μεταφορά σίγουρα είναι βασική πηγή τη ατμοσφαιρική ρήπανση. Θα πρέπει λοιπόν να αναζητήσουμε λύσει ώστε να περιορίσουμε τέτοιε μεταφορέ σε τόσο μεγάλε αποστάσει, ώστε να μην συμφέρουν πια τέτοιε μεταφορέ. Θα πρέπει να βρεθούν κάποιε οικονομικέ λύσει, ώστε να καταστούν πλέον μη προσοδοφόρες οι μεταφορές σε τόσο μεγάλες αποστάσεις ζώων. Γιατί όσο και αν προσπαθεί κανεί να εξασφαλίσει καλέ συνθήκε μεταφορέ, αν μιλούμε για μεταφορέ χιλιάδων χιλιόμετρων, είναι αδύνατον να είναι καλέ οι συνθήκε. Θα πρέπει λοιπόν να βρεθούν τρόποι να περιοριστούν ή να εξαλειφθούν αυτέ οι μεταφορέ σε τόσο μεγάλε αποστάσει. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και την ευκαιρία που μα δώσατε να σας παρουσιάσουμε την ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου στην Επιτροπή σας. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε κύριε Βοητσοχόφσκι εκ μέρους των μελών της Επιτροπής Γεωργίας. Σας ευχαριστούμε για την ε, παρουσίαση αυτής της πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση του Ελεκτικού Συνεδρίου. Όπως σας είπα, έχουμε τρία σημεία που αφορούν την καλή διαβίωση, την καλή μεταχείριση των ζώων. Είχαμε πρώτα την παρουσίαση της ειδική έκθεση του Ελεκτικού Συνεδρίου με θέμα την καλή μεταχείριση των ζώων. Τώρα θα ακούσουμε την παρουσίαση μιας μελέτης ε, του, της Υπηρεσίας Μελετών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον κανονισμό υπαριθμών 1 του 2005 για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά και τις συναφείς δραστηριότητε. Πρόκειται για το σημείο 7 δηλαδή της σας διάταξης, αλλά και το σημείο 8 είναι παρεμφερές γιατί αφορά την έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού 1 του 2005, την έκθεση Dorman. Περνάμε λοιπόν στο σημείο 7 τώρα, την παρουσίαση της μελέτης της Υπηρεσίας Μελετών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον κανονισμό 1 του 2005. Αποχαιρετούμε τον κύριο Βατσεχόφσκι και τον ευχαριστούμε για την καλοσύνη που είχε να έρθει στην Επιτροπή. Και περνάμε αμέσως στο σημείο 7. Όπως ξέρετε, για το σημείο 7, η διάσκεψη των Προέδρων σύστησε στην Επιτροπή μας την εκπόνηση μιας μελέτης εφαρμογής ε, για να εξακριβωθούν η κακή διαχείριση και οι πιθανές ε, ατασταλίες σε ό,τι αφορά το, την εφαρμογή του κανονισμού 1 του 2005 για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά. Σήμερα θα ακούσουμε την παρουσίαση δύο μελετών που αξιολογούν την εφαρμογή του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μεταφορά των ζών. Επίσης, η παρουσίαση αυτή, όπως σας είπα, σχετίζεται άμεσα με την έκθεση του κυρίου Ντόρμαν, που είναι το αντικείμενο της, το επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, το σημείο 8. Οι δύο μελέτες που θα μας παρουσιάσουν οι καλεσμένοι μας εκπονήθηκαν από την Υπηρεσία Μελετών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η πρώτη μελέτη είχε το, τον τίτλο ε, «Εφαρμογή του κανονισμού 1 του 2005 για την περίοδο ε, μέχρι το 2015 με βάση το Μητρό Δεδομένων». Δύο είναι οι συντάκτες της έκθεσης, ο κύριος Μπαλ, Μπάλτουσεν και ο κύριος Βάγκεμπερκ από το οικονομικό κέντρο, το ερευνητικό οικονομικό κέντρο του Wageningen από τις κατοχώρε. Δεύτερη έκθεση αφορά την εφαρμογή των τεχνικών κανόνων για την κατάλληλη φυσική κατάσταση των ζώων προς μεταφορά, όπως προβλέπει το παράρτημα 1 του κανονισμού 1 του 2005 για τη μεταφορά των ζώων κατά τη... για τη μεταφορά των ζώων, για την κατάσταση των ζώων κατά τη μεταφορά. Και εδώ έχουμε δύο συντάκτες της μελέτης, τον κύριο Βαν Σπόσλερ και τον κύριο Όγκεμπερτ. Πάλι από το Πανεπιστήμιο Βαγγενίγκεν, το ερευνητικό κέντρο της χώρα, της, των κατοχωρών. Θα ήθελα λοιπόν να καλωσορίσω τον κύριο Μπάλτουσεν, που είναι συνεισηγητής της πρώτης μελέτης Κύριε Βάλτους, αν έχετε ένα τέταρτο, μπορείτε να μας παρουσιάσετε μόνος ή με τον συνάδελφό σας τη μελέτη. Θα ακολουθήσει γύρω με ερωταπαντήσεις, ως συνήθως. Αλλά πρώτα να δώσω στο λόγο στην κυρία Λίνα Αντίνου, της Υπηρεσίας Μελετών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για μια σύντομη παρουσίαση αυτής της μελέτης για την εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας του κανονισμού 1. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Αξιότιμα μέλη. Με χαρά σας παρουσιάζουμε σήμερα την αξιολόγηση εφαρμογής πριν από τους ειδικού της έρευνας του Παγγενίγκεν. Και θα ήθελα με την ευκαιρία να πω πως η μονάδα μου έχει κάνει 61 εκ των υστέρων αξιολογήσει στην τρέχουσα βουλευτική θητεία, αλλά αυτή είναι η πρώτη για την Επιτροπή σας. Ελπίζουμε έτσι να ξεκινήσει και μια όμορφη φιλία που θα συνεχιστεί και στο μέλλον. Μερικά στοιχεία μόνο για να ξεκινήσουμε δεν μπορέσαμε να προβούμε σε μια πλήρη αξιολόγηση του κανονισμού για τους λόγους που ε, εξηγούμε στο εισαγωγικό τμήμα. Πάντως, και βάσει των στοιχείων που κοιτάξαμε, καταλήξαμε πως ε, η εφαρμογή παρουσιάζει μια ανάμεικτη εικόνα και με πρόοδους αλλά και με σημεία που σημειώνονται ακόμη προβλήματα αλλά και πραγματικές ανησυχίες και μελήματα όλων των εμπλεκομένων φορέων που έχουν ε, πάντα να κάνουν με την εφαρμογή. Τελευταίο, αυτή η αξιολόγηση έχει να κάνει με έρευνα από το γραφείο, δηλαδή δεν έχουμε συλλέξει νέα στοιχεία για την αξιολόγηση αυτή, όπως είπε ήδη ο Πρόεδρος, ο κ. Μπάρτουσεκ. Μπάλτουσεν της Balgeningen ε, Economic Research σας κάνει μια λεπτομερέστερη παρουσίαση των δύο εκθέσεων και σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Αντίνου και δίνω μέσω στο λόγο στον κύριο Μπάλτουσεν. 15 λεπτά. Πρόεδρε, ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Θα φροντίσω να μην ξεπεράσω τα 15 λεπτά. Πολλά εκατομμύρια ζώα ε, μεταφέρονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε μεγάλες αποστάσεις κάθε χρόνο. Αυτός είναι ο τομέας των μεταφορών των ζώων και άλλωστε είναι και ο λόγος για τον οποίο εισήχθη ο κανονισμός ΕΣΥ 1-2005 και ισχύει από το 2005. Αναφέρθηκε και νωρίτερα ότι η αξιολόγηση δεν είναι πλήρης. Περιοριζόμαστε λοιπόν σε συγκεκριμένα θέματα, θα σας εξηγήσω στη συνέχεια πια. Και ξεκινώντας, θέλω να πω ότι αυτή η μελέτη από γραφείου στηρίζεται στη φιλολογία, την τα επιστημονικά συγγράμματα δηλαδή, τα εφιστάμενα δεδομένα που έχουμε για την μεταφορά ζώων και από τα γραφεία τροφίμων και υπηρεσιών, από τα κράτη-μέλη και το και ορισμένες ολίγες συνεντεύξεις που έχουμε διεξαγάγει. Περίοδος μελέτης 2009-2015. και ουσιαστικά αφορά τα δύο πρώτα χρόνια υλοποίηση του κανονισμού. Άρα, στην περίοδο εκείνη που γινόταν η μελέτη, δεν είχαμε πολλά δεδομένα στη διάθεσή μα, ήδη δηλαδή το 2015. Πεδία εφαρμογή. Μόνο ζώα εκτροφή Δεν κάναμε δηλαδή έρευνα ε, για τα ζώα, για τα ζώα και ούτε για τα ζώα συντροφιάς. Η γενική εφαρμογή στα κράτη-μέλη είναι τα θέματα που εξετάσαμε. Τα, οι φορτωτικές και η διάρκεια του ταξιδιού, όπως δηλώνεται, η τήρηση του κανονισμού, η εφαρμογή, επιβολή του κανονισμού δηλαδή και η συμμόρφωση. γενική τήρηση των όρων του κανονισμού. Πέντε είναι τα σταθερά κριτήρια. Συνάφεια. Εάν παραμένει σημαντικός δηλαδή και έχει συνάφεια αυτός ο κανονισμός, ναι βεβαίως, γιατί ε, αυξάνεται διαρκώς ο τομέας των μεταφορών ζών των ζώων σε διεθνές επίπεδο, των διεθνών μεταφορών συγκεκριμένα. Αποτελεσματικότητα, δύσκολο να αναλυθεί η αποτελεσματικότητα, γιατί δεν έχουμε άξιόπιστους δείκτες για την ευημερία των ζώων. Άρα μπορούμε να κάνουμε κάποια σχόλια για τις συνθήκες της μεταφοράς, αλλά για τις συνέπειες τους και την ουσία της έρευνας που είναι η ευημερία των ζώων. Δεν μπορούμε. Αποδοτικότητα. Δεν είχαμε εναλλακτική. Άρα δεν μπορούμε και να ελέγξουμε πόσο αποδοτικός είναι ο κανονισμός σε σχέση με κάποιον άλλον που ενδεχομένω να υπήρχε. Συνοχή τα κύρια προβλήματα έχουν να κάνουν με τους χρόνους οδήγησης και ανάπαυση των οδηγών. Και έχουμε νομολογία του δικαστηρίου πλέον που μας λέει ότι είναι υποχρεωτικό η ώρα ανάπαυσης να πραγματοποιείται την ώρα που πρέπει να ξεκουραστεί ο οδηγός, ακόμα και αν αυτό σημαίνει ότι το ταξίδι, το δρομολόγιο θα παραταθεί και άρα θα μείνουν πιο πολύ ώρα στο ταξίδι τα ζώα η προσθέμενη αξία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι προφανή. Το πρώτο θέμα λοιπόν που έχει να κάνει με την καταγραφή των δρομολογίων με βάση και τις εκθέσεις των γραφείων τροφίμων και κτηνιατρικών θεμάτων. Βλέπουμε να βελτιώνεται η απόδοση, ωστόσο είναι σημαντικές αποκλήσεις μεταξύ κρατών μελών ακόμη. οι διαφορές έχουν να κάνουν και με το πόσα είναι τα δρομολόγια που καταγράφονται και με τη δράση που θα αναλυφθεί σε περίπτωση παράβασης και με τις ενδεχόμενες κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. Όλα αυτά τα θέματα λοιπόν παρουσιάζουν ε, αποκλείσεις μεταξύ κρατών μελών. Επιβολή του κανονισμού, επιβολή της εφαρμογής 1.2005 με κύριες πηγές ε, της δηλώσεις των κρατών μελών και των αντίστοιχων κτηνιατρικών ε, υπηρεσιών, υπηρεσιών ε, γραφείων τροφίμων. Βλέπουμε διαφορές. Βλέπουμε να βελτιώνεται η εναρμόνιση όμως παρόλα αυτά. Βλέπουμε να υπάρχουν ακόμη μεγάλες διαφορές στις κυρώσεις, σε περίπτωση μη Βελτίωση τη στήριξη των όρων του κανονισμού με την ανταλλαγή βέλτιστων των πρακτικών επίση σημειώνεται. Και από την τεκμηρίωση και τις συστάσεις της ΕΦΣΑ που είδαμε, δεν μπορούμε να καταλήξουμε εάν αυτές οι συστάσεις οδηγούν ή μπορούν, έχουν δυναμικό να οδηγήσουν σε ενίσχυση της ευημερίας των ζώων καθώς δεν μπορούμε να μετρήσουμε την ευημερία των ζώων, αφού δεν έχουμε δείκτες. Το τέταρτο στοιχείο που μελετήσαμε, καταλληλότητα για τις μεταφορές, καλή κατάσταση, ενός ζώου. Τι σημαίνει αυτό, ότι πρέπει να είναι υγιές το ζώο, την ώρα που θα φορτωθεί για να μεταφερθεί. Για να μπορέσει να αντέξει την, υπονόμε, την μείωση της ευημερίας την ώρα της μεταφοράς. Άρα κάθε ζώο πρέπει να ελέγχεται πριν την ε, φόρτωσή του ως προς την καταλληλότητα και αυτό με διαφορούς παράγοντες οι οποίοι έχουν την ευθύνη στη μεταφορά των ζώων ή απόδευους. για να προχωρήσω πιο γρήγορα. Καταγράφουμε τα συστήματα τήρησης των όρων του κανονισμού για τα δύο έτη 2014-2015, όπως μας τα καταγράψαν τα κράτη-μέλη, με το σύστημα το εναρμονισμένο καταχώρησης ε, της ε, παράβασης των όρων του κανονισμού. Και εδώ έχουμε, στον πίνακα αυτών, ποσοστά υψηλότερα όλων ε, σε θέματα παράβαση των όρων του κανονισμού ως προς την καταλληλότητα των ζώων για τις μεταφορές 2014-28% του συνόλου των παραβάσεων και 43% ακόμη περισσότερο το 2015. 43%. Υψηλά ποσοστά στην παραβίαση των όρων είχαν να κάνουν με τις πρακτικές των μεταφορών, το ύψος και τον, ε, τους χώρους ε, των φορτηγών κτλ. Κύριε Βρέματα, τεράστιες διαφορές, όπως είπα και πριν, μεταξύ κρατών σε σχέση με τον αριθμό των επιθεωρήσεων, από 0 έως εκατομμύρια υποθεωρείς τον χρόνο και αντίστοιχα παραβάσεις καταγραφόμενες από τα κράτη-μέλη και καταχωριζόμενες που μπορεί να είναι μηδέν για ορισμένα κράτη, μηδέν παραβιάσεις μέχρι και 7%. Και βέβαια σε αυτά τα κράτη που έχουν μηδενικέ παραβάσει, μηδενικέ είναι, μηδενικές είναι και επιθεωρήσει γιατί δεν έχουν αλλάξει τίποτα και άρα δεν έχουν βρει καμία παράβαση. Έχουμε 0 έως 7% λοιπόν καταχωρήσεις παράβασης των όρων του κανονισμού με μία εξαίρεση 16,6% την Ιρλανδία που, ε, που, έλεγξε και βρήκε 16% παραβάσεις. Τα πουλερικά είναι και που ελέγχονται το συγχρονότερο στα 2 αυτά χρόνια. Και οι συχνότερες παραβάσεις των όρων του κανονισμού καταγράφονται στην άφεξη στο σφαγείο. Στο άλλο ταξιδιού δηλαδή. Διαφορετικές στρατηγικές επιθεωρήσεων μεταξύ κρατών μελών έχουν επίσης καταγραφεί. Περισσότερες με βάση διακινδύνευση, ε, άλλες όχι. Εδώ βλέπουμε αποκλήσει και στον αριθμό των επιθεωρήσεων των ελέγχων και στην καταγραφή των παραβάσεων. πάνε από το 0 πάλι έως το 6%. 0 έως 5.000 επιθεωρήσεις ή έλεγχοι το χρόνο. Κύριε Ευρήματα, από τους ελέγχους επιτροπής. Από τους ελέγχους επιτροπής, λοιπόν, βλέπουμε ότι οι περισσότερες παραβάσεις έχουν να κάνουν με τους κανόνες περί των ζώνων μεταφορά. Πολλοί ε, επίσης παραβάσεις σχετίζονται και με τον τρόπο διάγνωσης της κοίησης, εφόσον αναφέρεται ξεκάθαρα το κανονισμό της ε, ύστερο της κοίησης δεν επιτρέπεται να μεταφέρεται τα ζώα. Κλήσεις βλέπουμε σε σχέση με το τι σημαίνει καταλληλότητα. Για παραδείγματα είναι τραυματισμένο να ζω βαρύ, βαρύς πρέπει να είναι αυτός ο τραυματισμός για να κρυθεί ακατάλληλο για μεταφορά. Πρακτικές αλλά και οικονομικές επίσης, ε, πρακτικά και οικονομικά κομμελήματα που μπορεί να έχουν ε, να κάνουν με την ε, διαπίστωση αν ένα ζώο είναι κατάλληλο ή όχι για μεταφορά. Και ένα ζήτημα που επανέρχεται πολλές φορές είναι τι συμβαίνει αν διαπιστωθεί ότι ένα ζώο δεν μπορεί να φορτωθεί για μεταφορά. με βάση την έρευνα και τα αποτελέσματα. Τα κράτη-μέλη πρέπει να ε, καταχωρίζουν ε, εναρμονισμένα δεδομένα για τις επιθεωρήσεις, τις μεταφορές και τις σχετικές, τις διαπιστωθήσεις παραβάσεις. Πρέπει να καταβληθούν επιπλέον προσπάθειες για να μειωθεί το επίπεδο παράβαση των του κανονισμού ή μη συμμόρφωσης. Έλεγχοι πρέπει να γίνονται περισσότεροι στο, στην καταλληλότητα κατά τη φόρτωση. Πρέπει να βελτιωθεί το σύστημα καταχωρήσεων σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης ε, για τα ζώα και τις ημερομηνίε γεννήσεως. Καλύτερη κατάρτιση χρειάζεται για οποιονδήποτε έχει να αναμειγνύεται στην ε, ευημερία των ζώων, ώστε να μπορούν καλύτερα να διαγνώσκουν την ακαταλληλότητα και αυτό αφορά όχι μόνο τον ε, κτηνοτρόφο αλλά και τους ε, υπαλλήλου που θα κάνουν τις επιθεωρήσεις. Ε, πρέπει να διαρευνούνται ε, οι εσδήποτε δυνατότητες υπάρχουν, να αποφεύγεται η μεταφορά των ζώων στο σφαγείο, αν υπάρχει δυνατότητα in situ σφαγής δηλαδή, και πρέπει να μειωθούν οποιαδήποτε οικονομικά κίνητρα μπορεί να υπάρχουν για τη μεταφορά ζώων σε πολύ μικρή ηλικία όταν αυτά είναι πιο ευάλωτα. Αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε μια συμφωνία κυρίων για την ενίσχυση της ευημερίας των ζώων κατά τις μεταφορές, συμφωνία κυρίων μεταξύ του κλάδου και των αρμοδίων αρχών, μπορεί να βελτιώσει οπωσδήποτε σημαντικά την Εφημερία των ζώων. Επίσης συνιστούμε ανταλλαγή πληροφοριών και γνώσεων για την ε, ε, βελτίωση της ευημερίας των ζώων με το σύστημα των των πρακτικών. Επί παραδείγματι, οδηγεί για το πώς πρέπει να γίνονται μεταφορές. Αυτό έχει αναπτυχθεί στη συνεργασία μεταξύ με κυβερνητικών οργανώσεων και μεταφορικών εταιριών βοήθησε μεταφορικές εταιρείε να αλλάξουν συμπεριφορά και να βελτιωθεί έτσι η ευημερία των ζώων. Ανταλλαγή πληροφοριών και γνώσεων μεταξύ και κρατών μελών. Παραδείγματι, με αποτέλεσμα την αναρμόνιση της, ε, του ελέγχου συμμόρφωση σε επίπεδο κρατών μελών. Σας ευχαριστώ θερμά για την προσοχή σας. χρόνο σας. Να δώσω τώρα το λόγο στον εισηγητή μας, τον κύριο Ντόρμαν. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, και σας ευχαριστώ για αυτά που μας είπατε ε, και τον τρόπο με τον οποίο μας περιγράψετε την κατάσταση και ως προς τα προβλήματα και ως την πρόοδο. Έχουμε αρκετές προκλήσεις να αντιμετωπίσουμε λόγω των μεγάλων διαφορών που υπάρχουν στα κράτη-μέλη. Αυτό που με προβληματίζει είναι υπάρχουν δυνατότητες για μια πιο ομοιόμορφη κατάσταση, μια εναρμόνιση ε, στον τρόπο μεταχείριση των ζώων για να αποφύγουμε την σημερινή κατάσταση όπου ουσιαστικά δίνουμε κίνητρα στις χώρες που δεν έχουν καλές να μεταφέρουν ζώα. Και μάλιστα όταν μεταφέρονται ζώα εκτός, εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περνούν ε, πολύ χρόνο στα σύνορα, σε ένα no man's Το θέμα είναι πώς θα επεξεργαστούμε τα στοιχεία που έχουμε για τις μεταφορές με βάση τις παραδοτικές και το χρόνο παράδοσης. Έχει γίνει κάποια πρόοδος, αλλά δυστυχώς πολύ περιορισμένη. Πόσο καιρό ακόμη πρέπει να περιμένουμε μέχρι ότου να εξασφαλίσουμε μια αξιοπρεπή μεταφορά των ζώων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ κυρία Νόιχλ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να φερθώ σε κάποια σημεία της παρουσίας, αλλά να συμπληρώσω και μερικά δικά μου Μιλήσατε για ελάχους, μιλήσατε για δεδομένα, είπατε ότι έχει χρησιμοποιήσει τα δεδομένα που ήταν στη διαθέση σας ήδη. Φαντάζομαι ότι είναι δεδομένα που καλύπτουν όλη την Ευρωπαϊκή Επικράτη, έτσι. Γιατί βλέπω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ακολουθεί μια σταθερή ε, τακτική αποφυγή των ελέγχων εκτός της επικράτειάς της. Δηλαδή δεν κάνουμε τίποτα μέχρι ότου φτάσει στον τελικό ε, προορισμό του το ζώο. Είτε είναι ε, αυτό στη Ρωσία, αυτός ο τελικός προορισμός, είτε είναι στο Ιράκ, έπρεπε κανονικά όλοι οι έλεγχοι να συνεχίζονται μέχρι το τελευταίο στάδιο του προορισμού. Ερωτώ λοιπόν εάν αυτοί οι έλεγχοι αφορούν μόνο την Ευρωπαϊκή Επικράτεια, εάν κάνετε και έλεγχου ε, όταν ε, τα ζώα βγαίνουν εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση. Μεταφερόμενα επίση, είπατε ότι μεγάλο κομμάτι των παραβάσεων ε, έχει να κάνει το 28% συγκεκριμένα με την καταλληλότερα για μεταφορά. Από το ένα μικρό ποσοστό των παραβάσεων που διαπιστώθηκαν είναι το 28% αυτές οι παραβάσει σχετικέ με, την, ε, με τον έλεγχο καταλληλότητα. Ήθελα λοιπόν να ρωτήσω εδώ έχει να κάνει αυτό το πρόβλημα με μια μεμονωμένη ατομική απόφαση που έχει λάβει κάποιο την ώρα που το ζώο πρόκειται να μεταφερθεί ε, και άρα δεν διαπιστώνεται ότι είναι κατάλληλο. Είναι και, γιατί εγώ αυτό βλέπω, διαρθρωτικές ε, διαρθρωτικά προβλήματα, παραβίαση δηλαδή των όρων καταλληλότητας, γιατί πρέπει όταν φτάνει ένας οδηγός φορτηγού να παραλάβει ζώα από το, εκμετάλλευση πρέπει να ξέρει αν θα, πάρει, αν θα παραλάβει ε, ή αν ε, θα παραλάβει πρόβατα. Αναλόγως θα είναι και το φορτηγό το οποίο θα οδηγήσει, με το οποίο θα πάει στην εκμετάλλευση. Αυτό υπάρχει, έχει πιστεί σαν πρόβλημα. Επίσης, Επίσης, αποτελεί απόλυτη ε, απόδειξη ανεπάρκειας και παινίας Ευρωπαϊκής Ένωσης το να είμαστε εξαρτημένοι από τη δουλειά που θα κάνουν μη κυβερνητικέ οργανώσει. Δηλαδή, εμεί δεν είμαστε, μην είμαστε σε θέση να επιβάλλουμε την νομοθεσία, αλλά να περιμένουμε από τι μη κυβερνητικέ οργανώσει να μα υποστηρίξουν. Βεβαίω να μα υποστηρίζουν, αλλά δεν είναι δυνατόν εξαρτώματα από τη δουλειά, εξαιρετική δουλειά το λέω βεβαίω ρητά, των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Και μια προσωπική παρατήρηση, το είπε και ο συνάδελφο νωρίτερα και σε μια άλλη έκθεση. Ε, έγινε λόγος για την ανάπτυξη πέθρου. Γιατί να μην γίνεται η σφαγή σε επίπεδο περιφερειακό, σε μικρά σφαγεία όπως συνέβαινε παλιά. Γιατί να έχουμε επικεντρωθεί, να γιατί να έχουμε συγκεντρώσει τη σφαγή σε μεγάλα μόνο σφαγεία και να πρέπει να γίνεται και η μεταφορά και να χάνεται και η συνάφεια με την περιοχή ολόκληρη την ε, περιφέρεια στην οποία βρίσκεται η εκμετάλλευση, γιατί τόσο πολύ επιμένει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη συγκέντρωση αυτή και γιατί να μην μπορούμε να αναλάβουμε δράση μέχρι και το σφαγείο στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο της μικρότερης περιοχής ή περιφέρειας. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα μας ε, έλυνε πάρα πολλά προβλήματα γιατί θα μπορούσε από τη μία μέρα στην άλλη με ένα μικρό δηλαδή, ταξίδι να μεταφερθεί το ζώο σε ένα σφαγείο ε, κοντινό ε, της ε, περιοχής για την σφαγή χωρίς. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ερώτημα. Είναι λογικό αυτό που κάνουμε τελικά. Ευχαριστώ. Κυρία Σράιερ, αλλά για δύο λεπτά παρακαλώ, γιατί πολύ χρόνο. Συγγνώμη που δεν πρόφερα καλά το όνομά σας, κυρία Σράιερ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Δεν είχα καταλάβει καν ότι ήρθε η σειρά μου. Μια σύντομη ερώτηση, αλλά σημαντική ερώτηση. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τους ομιλητές για τα όσα είπαν. Το πρόβλημα είναι η εφαρμογή της νομοθεσίας στην Ευρώπη. Είναι ανάγκη να το λύσουμε το ζήτημα αυτό. Αν έχουμε την κατάλληλη νομοθεσία θα πρέπει να υπάρχουν και οι ανάλογες κυρώσεις. Μπορείτε να πείτε κάτι παραπάνω γι' αυτό. Μιλάμε για τα οχήματα που δεν είναι κατάλληλα. Σε πολλές περιπτώσεις έχουμε 10 ώρες διαδρομής. Όταν δεν έχουμε το κατάλληλο όχημα είναι πρόβλημα όταν τα μισά από τα οχήματα δεν είναι όχι απλά κατάλληλα, σε καμία περίπτωση δεν προσεγγίζουν τις προϋποθέσεις. Σε ό,τι αφορά τα σφαγεία τώρα, θα ήθελα να πούμε κάτι παραπάνω και γι' αυτό. Όλα τα ζώα σφάζονται στα σφαγεία στη συνέχεια θα πρέπει να μεταφερθούν και από εκεί. Θα ήθελα να μάθω και παραπάνω για αυτά, γιατί και αυτό είναι ένα προβληματικό ζήτημα. Ευχαριστώ κύριε Χάζεκαμπ. Ευχαριστώ. Πιστεύω είναι κρίμα που είχατε τόσο λίγο χρόνο για να κάνετε την έρευνά σας. Και θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την τόσο καλή δουλειά που κάνατε παρά τα περιορισμένα μέσα που διαθέτετε και παρά τον περιορισμένο χρόνο που είχατε. Και διορθώστε με αν κάνω λάθος, επικεντρωθήκατε σε δύο σημεία κυρίως. Αναφερθήκατε στην καλή φυσική κατάσταση των ζώων και στα ζώα που προορίζονται για σφαγή. Σε ό,τι αφορά τη φυσική κατάσταση τώρα, έχω ένα ερώτημα. Είπατε ότι θα πρέπει να υπάρχουν περισσότερη έλεγχη στο σημείο άφηξης. Έχω περάσει κάποιο χρόνο στην Ανατολική Ευρώπη εξετάζοντας τις εξαγωγές των ζώων σε χώρες που βρίσκονται μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα ζώα φτάνουν υπερθερμανσμένα, ταλαιπωρημένα, εξαντλημένα, τραυματισμένα εξαιτίας των συνθήκων μεταφοράς ακόμη και αν είναι σε πολύ καλή φυσική κατάσταση μετά από μία-δύο ημέρες ταξιδιού μεταφοράς, αλλάζει τελείως η φυσική τους κατάσταση. Πώς μπορούμε να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Και με μία σειρά από μη καπαόμικρον. Έχω δει αρκετές ελλείψεις σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας. Δεν υπάρχουν έγγραφα που να ελέγχονται, δεν υπάρχουν κτηνίατροι παρόντες και δεν υπάρχει κανένα σύστημα επιβολής κυρώσεων. Επομένως, δεν υπάρχει τρόπος να, να δράσουμε σε περίπτωση παραβάσεων. Αυτό δεν αναφέρεται στην ε, έκθεσή σας και δεν κάναμε λόγο καν και για τη διαφθορά. Σε πολλές φορές βλέπουμε ότι είναι όλα καλά τυπικά. <clears throat> Ναι, ευχαριστώ πολύ για την έκθεση. Και βεβαίω η ερώτηση, κύριε, είναι γιατί να μεταφέρονται τόσο πολλά ε, ζώα σε τέτοιε αποστάσει στην Ευρώπη. Γιατί και μόνο γιατί είναι χαμηλότερο το κόστος το, από το ένα σφαγείο σε ένα άλλο. Εάν γίνεται αυτό, εάν συμβαίνει να είναι χαμηλότερο το κόστος από το ένα σφαγείο σε κάποιο άλλο, οφείλεται όμως στο ότι υπάρχουν τελείως διαφορετικές συνθήκες κοινωνικές, μισθολογικές κτλ. Και έτσι είναι ένας αθέμητο ανταγωνισμός αυτός που φέρνει χαμηλότερο κόστος και άρα την ανάγκη για τις μεταφορές των ζώνων. Έλεγχοι, επιθεωρήσεις. Γίνονται, πόσο γίνονται. Όταν έχουμε ποσοστό 0 στις επιθεωρήσεις, προφανώς δεν μπορούμε να ε, επιβάλλουμε τους ελέγχους, αλλά υπάρχει κάποιο είδους εποπτεία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να λέει στα κράτη-μέλη κάποιες προδιαγραφές στους ελέγχους πρέπει να τις έχετε και είναι αυτές και αυτές. Γιατί δεν νομίζω ότι κανένα κάνας μέλο θέλει να κάνει ε, δυσμενεί εκθέσει για τον εαυτό του. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν σχετικέ ε, αρχές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που επιβλέπουν τον τρόπο διεξαγωγής των ελέγχων των επιθεωρήσεων δυνατότητα για σφαγή στην ε, εγγύς περιφέρεια και περιοχή. Ναι, αλλά ούτως ή άλλως δυσκολίες υπάρχουν. Μπορεί η πιο συμπονετική για τα ζώα ε, σφαγή, ο πιο πολιτικός για τα ζώα τρόπος σφαγής να είναι στο λιβάδι, αλλά βεβαίως αυτό γεννά άλλες δυσκολίες. Δεν είναι εύκολο να βρίσκονται οι ε, συνθήκες εκείνες που επιτρέπουν την ε, η σωστή διαδικασία σφαγή κτλ. Και άρα ούτε αυτό μπορούμε να το επιτύχουμε. Για τι μη κυβερνητικέ οργανώσει, Θα πω και εγώ ότι αν οι μη κυβερνητικέ οργανώσει είναι αυτές που εξασφαλίζουν την τήρηση των προδιαγραφών και των κανονισμών στην Ευρώπη, είναι κακό δείγμα. Πρέπει λοιπόν να κοιτάξουμε κι εμεί από πλευρά μα πώ μπορούμε εμεί, οι βουλευτέ, κάποιοι άλλοι ενδεχομένω, να ασκήσουμε πίεση έτσι ώστε να προχωρήσουν αυτά τα θέματα, να μην περνούν μόνο από τι μη Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, κατακλείζομαι ηλεκτρονικά μηνύματα για τα προβλήματα με τις μεταφορές των ζώων. Η κοινή γνώμη ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τις συνθήκες μεταφοράς των ζώων. Θα πρέπει λοιπόν να διαχωρίσουμε δύο θέματα. Καταρχήν έχουμε τη μεταφορά ζώων και έχουμε και εισαγωγές και εξαγωγές ε, ζώων για σφαγή. Θα πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ρυθμίσει τις μεταφορές των ζωντανών ζώων προκειμένου να ενταχθούν σε προγράμματα αναπαραγωγής. Γιατί μεταφορά ζώων αναπαραγωγής δηλαδή. Όταν εγώ αγοράζω ζώα από οποιαδήποτε χώρα, από την Δυτική Ευρώπη για παράδειγμα, και τα εισάγω στη Ρουμανία, θέλω να είμαι βέβαιος τα ζώα αυτά είναι σε εξαίρετη φυσική κατάσταση όταν έρχονται στη Ρουμανία. Είτε χρησιμοποιούνται για αναπαραγωγή, είτε όχι. Άλλο όμω ε, όταν μιλάμε για ζώα ε, που έχουν ήδη σφαγεία, σφάγια, για μεταφορά σφαγείων. Υπάρχουν χώρε που έχουν περισσότερα σφαγεία ή πολύ κοντά στου τόπου εκτροφή. Ενώ άλλε χώρε δεν έχουν σφαγεία κοντά στι κτηνοτροφικέ μονάδε και χρειάζεται να μεταφερθούν τα ζώα είμαι σύμφωνος με την ανάγκη να παραμείνουν τα έσοδα σε μια περιοχή, να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης και να είναι βραχίες οι αλυσίδες. Αλλά τα ζώα πρώτα απ' όλα, όταν πηγαίνουν για σφαγή, θα πρέπει να είναι σε άριστη φυσική κατάσταση. Και πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει την ικανότητα και τη δυνατότητα να συνάψει συμβάσει με χώρες προορισμού για να ε, όταν έχουμε εισαγωγή από Ισραήλ, προϋποθέσεις προποθέσει τελετουργική φαγή. Είναι απαράδεκτο απ' την άλλη να εισάγουμε ζωντανά ζώα που μεταφέρονται σε πολύ μεγάλε αποστάσει και μετά από πολλή ώρα ταξίδια. Η ποιότητα του κρέατος, άλλωστε επηρεάζεται από τι συνθήκε μεταφορά. Όλα αυτά είναι σημαντικά. Ευχαριστώ κύριε Ριμπέιρο. σχόλιο για τις ε, μεταφορές των ζώων, γιατί είμαι σκιώδης συγγήτρια ε, της έκθεσης Dorman Θα ακολουθήσει όμως η συζήτηση αυτή γίνει και αργότερα. Θα ήθελα να θέσω μια συγκεκριμένη ερώτηση. Στη νέα έκθεση έχουμε διάκριση μεταξύ της ευθύνης του κτηνοτρόφου από την ευθύνη του μεταφορέα. Γιατί πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνει αυτή η διάκριση στην ευθύνη των δύο, κτηνοτρόφου και μεταφορέα. Γιατί τα συμφέροντά τους είναι πολύ διαφορετικά ο κτηνοτρόφος έχει κάθε συμφέρον να εξασφαλίσει την ε, μεταφορά με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες προκειμένου να φτάσει σε άριστη κατάσταση το ζώο στον, τρόπο, προορισμού. Αυτό τον ενδιαφέρει για τη δουλειά του. Γιατί όσο, σε όσο καλύτερη κατάσταση ε, φτάνει το ζώο, τόσο μεγαλύτερο θα είναι το κέρδος του κτηνοτρόφου οι μεταφορικές εταιρείες το μόνο που θέλουν είναι να εξασφαλίσουν τη μεταφορά άσχετα με τις συνθήκες της μεταφοράς. Έγινε διάκριση μεταξύ της ευθύνης του κτηνοτρόφου και της ευθύνης του μεταφορέα και αν ναι, τι συμπεράσματα προέκυψαν από, μια, από ένα τέτοιο διαχωρισμό των ευθυνών, γιατί είναι και διαφορετικά τα συμφέροντα. Ευχαριστώ κύριε Μαγκίνες. Um, Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστούμε και για την παρουσίαση. Σε ό,τι αφορά τους τραυματισμούς των ζώων που μπορεί να τραυματιστούν στα κτηνοτροφία, να σπάσουν ένα πόδι για παράδειγμα. Αυτό ξέρω ότι είναι ένα πρόβλημα που υπάρχει στη δική μου την περιφέρεια. Πρώτα απ' όλα ένα πρόβλημα ζώου μπορεί να είναι πολύ σημαντικό. Αν το ζώο αυτό δεν θεωρείται ότι είναι σε καλή φυσική κατάσταση για να μπορέσει να μεταφερθεί και δεν υπάρχει δυνατότητα να σφαγεί στο κτηνοτροφείο, και όντω σε πολλέ περιπτώσει το ζώο μπορεί να μην είναι σε κατάσταση να σφαγεί και μπορεί να φτάσει στο σφαγείο και τελικά να μην καταλήξει να σφαγεί. Και ένα κατάλληλο κρέα να πάει ανεκμετάλλευτο. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Το δεύτερο που ήθελα να πω, αναφερθήκατε συγκεκριμένα στην Ιρλανδία. Ένα νούμερο 16% εγώ Είμαι από την Ιρλανδία και ξέρω ότι κάνουμε πάρα πολλούς ελέγχους. Ξέρω ότι είμαστε αυστηροί. Επομένως, τι κάνουμε, συγκρίνουμε διάφορα κράτη-μέλη και ψάχνουμε το ίδιο ποσοστό. Είπατε ότι σε πολλά κράτη-μέλη είδατε 0%. Ενώ στην Ιρλανδία 16%. Μήπως θα πρέπει να επισέλθουμε λίγο σε λεπτομέρειες. Εγώ πάντοτε πίστευα ότι το πρόβλημα είναι εφαρμογή, είναι τελείως τυχαία. Σε κάποια κρατημέλη εφαρμόζεται νομοθεσία, σε κάποια, σε κάποια άλλα όχι. Είναι ανάγκη να έχουμε καλύτερη εφαρμογή. Το δεύτερο, το τελευταίο σημείο που θέλω να θίξω έχει να κάνει με τα μεγάλα σφαγεία που αποτελούν τον κανόνα τώρα. Η εμπειρία όμω που είχαμε όλοι είναι ότι τα μικρά σφαγεία κλείσαν. Σε πολλές περιπτώσεις οι τοπικές αρχές για λόγους ασφαλείας τα έκλεισαν, γιατί απαιτούνταν τεράστιες επενδύσεις, ε, κάτι το οποίο δεν ήταν συμφέρον για τον κτηνοτρόφο. Μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Ε, με ενδιαφέρει πολύ να, να δω τι σκέφτεστε πάνω σε αυτό το ζήτημα. ένα πρώτο ζήτημα. Αν θέλουμε να ρυθμίσουμε αποτελεσματικά την, το ζήτημα της καλής κατάστασης των ζώων κατά τη μεταφορά, είναι ανάγκη να βοηθήσουμε, την, να χρηματοδοτήσουμε τη δημιουργία σφαγίων, άσχετα με το τι μέγεθος θα είναι τα σφαγεία αυτά, αλλά πιστεύω ότι αυτή είναι η πιο αποτελεσματική λύση. Θα ήθελα να σας πενθυμίσω τη μεταφορά των ζωντανών ζώων και οι καλές συνθήκες υγιεινής είναι πάρα πολύ σημαντικές ε, για να μην σας υπενθυμίσω τις διάφορες επιδημίες που έχουμε διαπιστώσει στη Ρουμανία, στην Ουγγαρία και στην Γαλλία, την ταχύτατη ανάπτυξη, η πάρα πολύ γρήγορη κινητοποίηση στη Γαλλία και ο εμβολιασμό ε, των ε, αγελάδων ενάντια στον ε, πυρετό αυτών των αγελάδων βοήθησε στο να αποφύγουμε τις επιδημίες αυτές. Για να μην έχουμε και τεράστιες απώλειες. Σε πολλές περιπτώσεις θα ήταν ανάγκη να κλείσουμε και την εξαγωγή σε διάφορες τρίτες χώρες. Η Επιτροπή για μια ακόμη φορά βασίζεται στο ελεύθερο εμπόριο για να μην εφαρμόσει τις αρχές που ισχύουν. Σε πολλές περιπτώσεις όμως αυτό βλάπτει τους κτηνοτρόφους στην Ευρώπη και σε πολλές περιπτώσεις περιορίζει και τις τρίτες χώρες, οι οποίες θέλουν και αυτές να εξάγουν σε εμά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πολύ ενδιαφέρουσα η μελέτη, που μας παρουσιάσατε. Να σταθώ σε κάτι που είπε η κυρία Νόεχλ για τα μικρά, για τα μικρά σφαγεία. Το είπε και η κυρία Μαγκίνες. Φαίνεται ότι ε, πρέπει να κλείσουν αν δεν έχουν συγκεκριμένες διαστάσεις. Στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας πάντως έχουμε ένα σύστημα που αφορά ένα ζήθο που παράγουμε και για να ε, επιζήσουν τα μικρά ζυθοποιία πληρώνουν μικρότερο φόρο. Ήταν 200.000 λίτρα το όριο για να χαρακτηριστεί ένα ζυθοποιό μικρό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μα έλεγε στην αρχή δεν μπορείτε να το κάνετε. Τελικά το κάναμε και λειτουργεί μια χαρά. Και ίσως για πρώτη φορά στην Ελλαδία έχουμε πια μικρά ζυθοποιία που είναι βιώσιμα. Γιατί δεν μπορούμε κάτι αντίστοιχο να κάνουμε με τα μικρά σφαγεία. Ε, να έχουμε ένα κατόφλι σε περίπτωση που βρίσκονται κάτω από τον τζίρο και τον όγκο να έχουν κάποια φορολογικά κίνητρα ελαφρύνσης. Το ίδιο και για αρτοπία, γιατί ε, αν δεν έχουμε τέτοιες θετικέ θετικές ε, διατάξεις ε, για τέτοιου είδους ε, μικρά σφαγεία, αρτοπία κτλ. Δεν θα έχουμε στο τέλος στην, στην Ήπεθρο τέτοια επαγγέλματα και θα χρειαστεί να φύγουν όλοι προς τις πόλεις. Ενώ στην, στην Ιρλανδία τα καταφέραμε, αν μη τι άλλο, με τη την τοπική ζηθοποιία. Ευχαριστώ. τι τις μελέτες της Υπηρεσίας Μελετών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Συμφωνούμε σε μεγάλο βαθμό με τα πορίσματά της. Άλλωστε στηρίζονται οι μελέτες σε στοιχεία που έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το σύστημα TRACE, στο ενοποιημένο μηχανογραφικό κτηνιατρικό σύστημα που το διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και τα βασικά προβλήματα που εντόπισε η μελέτη είναι γνωστά όχι μόνο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και τους άμεσα ενδιαφερόμενους συνεργασία με τα κράτη-μέλη αναζητεί λύσεις στα προβλήματα αυτά. Για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά την εξαγωγή των ζώων και το πρόβλημα με τις θερμοκρασίες. Αυτό είναι ένα θέμα που αναφέρθηκε στις μελέτες. Μερικές χώρες από πέρυσι το καλοκαίρι απαγόρευσαν την εξαγωγή ζωντανών ζώων στην Νότια Ευρώπη. Και αυτό έγινε όπως πρότεινε η μελέτη από συμφωνίες των αρμοδίων αρχών. Οι αρμόδιες αρχές να μην ε, γίνονται μεταφορές όταν η θερμοκρασία ξεπερνά τους 30 βαθμούς. Έχουμε την Ιρλανδία, την Αυστρία, τη Γαλλία, τις κάτω χώρες που επίσης περιορίζουν τις εξαγωγές πάνω από μια θερμοκρασία. Επίσης, για μερικά προβλήματα οι λύσεις δεν είναι εύκολες. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να βρουν σε εθνικό επίπεδο Οπότε τα κράτη-μέλη είναι αυτά που θα πρέπει να εφαρμόσουν την νομοθεσία. Και καλώς ή κακώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να πεντάλεπτο για να επιχειρήσετε κάποιες απαντήσεις και μην κοιτάτε ε, με βλωσιρότητα. Έχουμε πολλά ακόμη σημεία στην ημερήσια διάταξη. Λυπάμαι που σας περιορίζω τόσο, γιατί είναι περίπλοκο το θέμα δεδομένης πληθώρας των ερωτήσεων, αλλά δυστυχώς λίγο χρόνο έχουμε. Έχετε το λόγο κύριε Βάλτους. Ε, ε, Ευχαριστώ για τα πέντε λεπτά που μου δίνετε να απαντήσω σε όλα αυτά τα ερωτήματα. Το πρώτο πράγμα που θέλω να πω για τα σφαγεία, για τα μικρά ή για τα μεγάλα, η μεταφορά των ζώων δεν εξαρτάται από τα μεγάλα ή τα μικρά σφαγεία. Πολλά ζώα μεταφέρονται από τις κάτω χώρες στη Γερμανία για να σφαγούν. Και τα ζώα αυτά ταξιδεύουν για μία-δύο ώρες. Και αν εξετάσουμε την περιοχή του Βελγίου και των κατοχωρών, γενικά υπάρχει πολλή μετακίνηση, η οποία είναι σύντομη μετακίνηση ζώων. Και αυτό γιατί είναι οικονομικά συμφέρον στη Γερμανία να σφαγούν τα ζώα εκεί. Και αυτό είναι μια απάντηση και σε ένα από τα ερωτήματα. Γιατί τόσα πολλά ζώα μεταφέρονται. Αυτό έχει να κάνει και με τις διαφορές ανάμεσα στις διάφορες περιοχές στην Ευρώπη που έχουν να κάνουν με την παραγωγή και την κατανάλωση. Αν καταναλώνεται περισσότερο κρέας σε ένα σημείο, σε μια περιοχή της Ευρώπης, τότε είναι λογικό να υπάρχει μεταφορά κρέατος ή και ζωντανών. Σε αρκετές δημοσιεύσεις έχουμε καταδείξει ότι η μεταφορά του κρέατος είναι πιο φτηνή από την μεταφορά ζωντανών ζώων. Παρ' όλα αυτά όμως, σε κάποιες περιπτώσεις προτιμούν οι άνθρωποι να μεταφέρουν ζωντανά. Επομένως, τα ζώα μεταφέρονται από τη μία περιοχή στην άλλη. Σε κάποια άλλη έκθεση είχαμε δείξει ότι ας πούμε πρόβατα από την Ουγγαρία μεταφέρονται στην Ιταλία και αυτό γιατί δεν υπάρχουν σφαγεία για πρόβατα στην Ουγγαρία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 μπορεί κανείς να τα σκοτώσει τα ζώα αυτά. Και μπορεί να είναι κατάλληλα για κατανάλωση στη συνέχεια. Ή μπορεί και να δοθεί η έγκριση να μεταφερθούν τα ζώα αυτά στα σφαγεία και το κρέας του στη συνέχεια να είναι διαθέσιμο για κατανάλωση. Για όλες αυτές τις επιλογές υπάρχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Το εξετάσαμε το ζήτημα αυτό, αλλά δεν έχουμε μια σαφή απάντηση αυτή τη στιγμή. Υπήρχαν επίσης ερωτήματα σχετικά με διάφορα κράτη-μέλη. Και με αυτό το οποίο είπα συχνά, ότι υπάρχουν πολλές διαφορές ανάμεσα στα διάφορα κράτη-μέλη. τουλάχιστον εν μέρει στα νομικά συστήματα που ισχύουν, αλλά και στις προτεραιότητες που υπάρχουν σε ό,τι αφορά την μη συμμόρφωση, σε ό,τι αφορά τις παραβάσεις, σε ό,τι αφορά τα πρόστιμα. Οι διαφορές αυτές επίσης είναι ένα ζήτημα που θα πρέπει να εξετάσουμε. Δεν κάναμε διάκριση μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών, γιατί δεν έχουμε συγκεκριμένες πληροφορίες από την έρευνά μας, επομένως δεν κοιτάξαμε τους κτηνοτρόφους ή τους μεταφορείς ή τους επίσημους κτηνίατρους κτλ. κτλ. Σε ό,τι αφορά την κοινή γνώμη τώρα, υπάρχει συζήτηση σε ό,τι τη μεταφορά των ζώων. Υπάρχουν φήμες και βλέπουμε, διαπιστώνουμε και καλές πρακτικές. Αν εξετάσουμε ειδικέ συνθήκες, όπως είναι ας πούμε, τα σύνορα Βουλγαρίας Τουρκία θα δείτε ότι δεν υπάρχουν καταγγελίες μισή και οι συνθήκες δεν είναι καλές, δεν είναι ευνοϊκές. περιμένει για 6 ώρες ακόμη και αν όλα πάνε σύμφωνα με το πρόγραμμα. Δεν είναι κάτι το θετικό αυτό, αλλά έτσι έχουν τα πράγματα. Σε ό,τι αφορά τώρα την καλή μεταχείριση των ζώων, είναι κάτι που δεν εξετάσαμε στην έρευνα αυτή και δεν γνωρίζω κατά πόσο είναι μεγάλο ο κίνδυνο. Βεβαιώς και υπάρχει κίνδυνο. Αν φέρει κανεί στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό χώρο, υπάρχει κίνδυνο ασθενειών μπορεί να έχουν να κάνουν με τη μετακίνηση. Δεν ξέρω όμως να σας πω πόσο εκτεταμένος είναι ο κίνδυνος αυτός. Χαίρομαι που καταφέραμε να περιλάβουμε στην έρευνά μας τις πληροφορίες που έχει ήδη η Επιτροπή, κάτι το οποίο κάναμε με τρόπο θετικό, όπως μας είπαν. Σε ό,τι αφορά τώρα που έχουν να κάνουν με τις συμφωνίες. Πιστεύω ότι στις κάτω χώρες πάνε και ένα βήμα παραπάνω. Λένε ότι αν η θερμοκρασία α, ξεπεράσει τους 30 βαθμούς, τότε δεν υπάρχει μετακίνηση. Αυτοί λένε επιπλέον ότι τον Ιούλιο και τον Αύγουστο δεν κάνουμε μεταφορές προς την Τουρκία. Επομένως, αυτή είναι ένα βήμα παραπάνω από την εφαρμογή του κανονισμού. Και αυτή η επιλογή υπάρχει. Και άλλες χώρες παραδείγματα το, ακόμα και μέσα στην ίδια την ε, γεωργική, την εκμετάλλευση ή στο εγκύτερο δυνατό και περισσότερο αποτρεπτικό χαρακτήρα και όχι τόσο τιμωρητικό, γιατί συνήθως είναι οι ίδιοι που εξαπατούν. Θα πρέπει να έχουμε λοιπόν ε, ε, καλύτερες κυρώσεις. Επίσης, ό,τι αφορά τη μεταφορά άρρωστων ζώων, αυτό δεν σημαίνει ότι όλες οι μεταφορές είναι κακές. Το γεγονό ότι κάποια ζώα πεθαίνουν στις μεταφορές σημαίνει ότι πρέπει να καταργήσουμε τις μεταφορές των απαγορεύαμε τις μεταφορές σε περίπτωση θανάτου, θα έπρεπε να είχαμε καταργήσει οδικέ μεταφορές, γιατί εκεί υπάρχουν πάρα πολλά τροχαία χώρα. Σίγουρα και η μεταφορά των ζώων επιδέχεται βελτιώσει, αλλά σε καμία περίπτωση πρέπει να απαγορευτεί. Επίσης, ό,τι αφορά τι θαλάσσιες μεταφορέ, συνεργασία με τις χώρες, ε, τρίτες χώρες εισαγωγής ε, ζώων. Θέλουμε να φτάνουν το ζώα στον προορισμό τους ε, σε καλές συνθήκε και με καλές προϋποθέσεις μεταφοράς. Επίσης, θέλουμε καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών, αξιοποιώντας και τις υπάρχουσες τεχνολογίες. Γιατί θα πρέπει να γνωρίζουμε είναι, ποιος είναι ο τελικός πρέπει να πετούμε για τα ζώα καλύτερες συνθήκες από ό,τι για τη μεταφορά ενδιαφέρον τη κοινή γνώμη για τα θέματα αυτά. Επίση, καλύτερη επιθεωρήση τους τρέχοντες κανόνες και τις αποτελεσματικές κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης και όχι κατά ανάγκη επισκεφθεί τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να δω την κατάσταση εκεί σε ό,τι αφορά τη μεταφορά των ζώων. Και όταν βλέπω τι συμβαίνει στην Κροατία και αλλού, πραγματικά οι συνθήκες αυτές δεν θα έπρεπε να, να τις ήταν ιδιαίτερα υψηλή. Τα ζώα ήταν τραυματισμένα, ήταν άρρωστα, ήταν υπερθερμανισμένα. Υπήρχαν κτηνίατρικοι, ήταν σαφές. Δεν υπήρχαν κτηνίατρικοι. Είναι σαφές ότι αν υπήρχαν εκεί θα προστάτευαν τη βιομηχανία. Και το χειρότερο, αυτό που είδα για πρώτη φορά το 1991 στη τηλεόραση και πάλι στην Κροατία, στο ίδιο λιμάνι, ήταν το ίδιο πράγμα. Ένα πλοίο το κρατούσαν από τα μπροστινά του πόδια και στη συνέχεια το χτύπησαν με ηλεκτρικές ράβδους για να προχωρήσει γιατί δεν μπορούσε να σταθεί στα πόδια του και δεν έγινε καταγγελία. Και αυτό είναι κάτι ανάλογο που βλέπουμε σήμερα στην Ευρώπη. Ακούσαμε εδώ θα μπορούσαμε να είμαστε λίγο πιο αυστηροί στη διατύπωσή μας. Η μετακίνηση, η μεταφορά των ζώων σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλοι λένε ότι είναι πολύ σημαντικό για τα ζώα να φτάσουν σε μια καλή κατάσταση. Αν ξέρετε τι συμβαίνει, να σας προτείνω ένα DVD που προβλήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στη Γερμανία, αν έχετε το στομάχι να μπορέσετε να το δείτε. Πραγματικά πρέπει να σταματήσουμε τις μεταφορές έξω από τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περισσότερα σφαγεία δεν θα μας λύσουν το πρόβλημά μας. Μία είναι των ζώων θα πρέπει να αλλάξουμε τις συνήθειες κατανάλωσης. Ευχαριστούμε και ότι για τους πράσινους. Ναι, ναι, νομίζω ότι έχουμε την ίδια συζήτηση πάντα και πάντα. Έκθεση. Αλλά ξαναρχόμαστε στο ίδιο ερώτημα. Είναι καλή η νομοθεσία μας. Και η απάντηση είναι, α, είναι καλύτερα από τους άλλους. Ναι, αλλά αυτό δεν είναι ε, η απάντηση, η τελευταία ανάλυση, πρέπει να έχουμε και σωστούς ελέγχους και σωστή εφαρμογή του κανονισμού που είναι καλύτερος από τους άλλους. Λοιπόν, καλό είναι να περιγράφουμε τα προβλήματα, αλλά δεν νομίζω ότι μπορούμε να περιοριστούμε μόνο σε αυτό, στο να περιγράφουμε τα προβλήματα. Και έστω να περιοριστούμε σε αυτό την πρώτη φορά, αλλά όχι κάθε φορά. Ένα εκατομμύριο υπογραφές συγκεντρώθηκαν που ζητούσαν οι πολίτες να τα αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό. Πρέπει λοιπόν να στήσουμε αυτή την Επιτροπή να αναλάβουμε στο το οποίο να μπορεί να επιβληθεί και με κυρώσεις, εάν δεν τηρείται. Διαφορετικά θα περιοριζόμαστε μόνο στο να περιγράφουμε το πρόβλημα, χωρίς όμως να το αντιμετωπίζουμε. Ε, το ζήτημα της ε, μείωσης του χρόνου των μεταφορών ή του περιορισμού του χρόνου των μεταφορών έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Το έχουμε συζητήσει επανειλημμένως. Γιατί να πρέπει να μεταφέρονται τα ζώα, το είπαμε και νωρίτερα, γιατί να πρέπει να διασχίσουν ολόκληρη την Ευρωπαϊκή η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί είναι φθηνότερα κάποια σφαγεία κάπου λόγω χαμηλότερων κοινωνικών προδιαγραφών. Μα αυτή η αυτές οι μεταφορές δεν θα έπρεπε να επιτρέπονται. Και έτσι το πρόβλημα δεν είναι να υποβαστούν τα σφαγεία παντού, αλλά να έχουμε πιο πολλά σε μικρή κλίμακα, σε ε, μικρότερες περιφέρειες σφαγεία που να μας είμαστε εμείς όσα απαιτούμε, είμαστε των όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση να εφαρμόσει, είναι μήνυμα νομίζω απαιτείται που αφορά και τις μεταφορές και τους ελέγχους και τις κυρώσεις. Αυτό θα είναι μια πραγματική προσθέμενη αξία. Οι τελετουργικές ε, σφαγές μπορούν να γίνονται από εδώ και μπρος, πρέπει να μπορούν να γίνονται από εδώ και μπρος μόνο συζήτηση δείχνει ξεκάθαρα ότι υπήρχε, υπήρχε να γίνει η συζήτηση αυτή και ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές σχετικά με το πώς εννοούν τις μετακινήσεις των ζώων τα διάφορα κράτη-μέλη. Πιστεύω ότι όλοι θα πρέπει να αποδεχτούμε ότι είναι αυτή η τεχνολογία που ισχύει τα τελευταία χρόνια και όταν μιλάμε για καλές φυσικές συνθήκες των ζώων, τότε θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας και τις αξιολογήσεις. Και οι αξιολογήσεις έχουν να κάνουν με το ποιος τις κάνει. Και βέβαια υπάρχει το ζήτημα συμμόρφωσης με τους κανόνες. Εγώ έχω διαπιστώσει μεγάλες διαφορές ό,τι αφορά την συμμόρφωση όπου υπάρχουν κυρώσεις. Μπορεί να βελτιωθεί η νομοθεσία. Βεβαίως και μπορεί και πιστεύω όλοι συμφωνούμε στο ότι καλύτερη δυνατή νομοθεσία, ούτως ώστε να μεταχειριζόμαστε τα ζώα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όταν μετοκινούνται. Είτε πρόκειται για την πρώτη, είτε πρόκειται για την τελευταία μεταφορά τους. Βεβαίως υπάρχουν διαφορές σχετικά με το αν αναφερόμαστε σε ζώα τα οποία πηγαίνουν στα εκτροφία ή σε ζώα που πηγαίνουν στα ασφαγεία. Αλλά πιστεύω ότι από κοινού μπορούμε να βελτιώσουμε καλή κατάσταση των ζώων και προσδοκώ την καλή μας συνεργασία. Ευχαριστώ. δομές του ε, επιπλέον κόστο που μπορεί να επιβαρύνει τον ε, ε, προμηθευτή. Ένα άλλο σημείο που έχει να κάνει με τη δυνατότητα να καταγγέλλεται μια παράβαση και από προμηθευτών, αυτό συμμερίζεται και η Αυστριακή Προεδρία, μάλιστα και από οργανώσει εκπροσώπηση και μη κυβερνητικέ οργανώσεις σε ε, αρκετά κράτη-μέλη, ακόμα και αν υπάρχει σχετική νομοθεσία, ελάχιστε προδιαγραφέ λοιπόν, και αυτό είναι ακόμα το οποίο έχει μπει στη διαπραγμάτευση. Ενσωμάτωση μηχανισμών μεσολάβηση και επίλυση διαφορών, όπω και στι επίση στο Κοινοβούλιο. Ενίσχυση τη συνεργασία μεταξύ όλων των εθνικών αρχών που επισχύστηκε στο Κοινοβούλιο. Εν γέννη, ε, βλέπουμε ότι αρκετά σημεία του Κοινοβουλίου κάνει με τη δυνατότητα της επέκτασης της εφαρμογής της οδηγίας σε κάθε προμηθευτή. Υπό την αρχή που όλοι χαιρετήσαμε με μεγάλο ενδιαφέρον, το unfair, unfair is unfair. Αθέμητο, το αθέμητο θα είναι πάντα αθέμητο και έτσι το Κοινοβούλιο δεν επιτρέπει, δεν θα δεχθεί κανένα περιορισμό στην εφαρμογή αυτής της αρχής. για να καταλήξουμε σε ένα συμβασμό. Το σημαντικό για μας είναι να εγκριθεί αυτή η σημαντική οδηγία, αλλά αναμένουμε και από την Αυστριακή Προεδρία, με βοήθεια βέβαια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κάποιες κινήσεις για τον τριμερή διάλογο της προσεχούς Πέμπτης, κάποια βήματα προόδου, που ωστόσο, Πρόεδρε, πρέπει να σημειώσω, μέχρι σήμερα δεν έχουμε δει. Και γι' αυτό και θα μια δυνατότητα διαμεσολάβησης προς την Αυστριακή Προεδρία έτσι ώστε να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ε, λύσεις σύμφωνες με αυτό που με ευρύτατη πλειοψηφία 328 υπέρ 170 κατά Είναι πολύ σημαντικό όμως να πούμε ότι πρόκειται για πολύ σημαντική νομοθεσία. Επομένως, προτιμώ να κάνουμε τα πράγματα σωστά παρά να βιαστούμε. Όλα τα μέλη της ομάδας θα εργαζόμενοι σκληρά και πέραν του ωραρίου τους. Υπάρχουν να κάνει μια έρευνα πάνω στο σημείο αυτό σε διαφορά την ε, νομοθεσία που έχουμε συμφωνήσει, καθώς επίσης και η τροπολογία 64 που δεν περιλαμβάνεται πλέον στο κείμενο. Αυτά θέλω να σας πολλά κάνει, έχουμε διαπραγματευτεί σκληρά, έχουμε επιτύχει πολλά και ιδιαίτερω χαίρομαι γιατί θα έχουμε τη δυνατότητα να ε, κερδίσουμε πολλά σημαντικά για τους παραγωγούς μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά έξω και από αυτή. Ε, και βέβαια αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να επεκταθεί και πέραν τη εξαρτάται ένας παραγωγός από το εμπόριο, αν ανήκει σε ένα συνεταιρισμό, αν είναι εκτεθειμένος στο ελεύθερο εμπόριο και εδώ νομίζω ότι χρειάζεται περαιτέρω προσπάθεια. Έχουμε δυσκολίες και στην αγορά και στην πώληση, την κάλυψη του κόστους ε, παραγωγής και γι' αυτό βλέπω ότι έχει μείνει μια γκρίζα ζώνη να τα κλείσουμε. Πρόκειται για έναν περισσότερο τεχνικό διάλογο, σημαντικό αυτό νομοθετικό σχέδιο. Η συνεργασία με την Αυστριακή Προεδρία ήταν επίσης επικοδομητική και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία στην τρέχουσα φάση του τριμερούς διαλόγου τη ε, τρέχουσας Εβδομάδα. Και θα ήθελα να υπογραμμίσω τα εξή. Πρώτον, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να δείξει ευελιξία και λογική ε, προσέγγιση όταν φτάσουμε στον προσδορισμό του πεδίου εφαρμογή τη οδηγία και τη χρήση διότι έχουμε μόνο για την εισαγωγή μέτρων που μπορεί να βελτιώσουν τις προδιαγραφές διαβίωσης των παραγωγών που μπορεί να είναι ο κύριος στόχος της οδηγίας αυτής και μόνο και πρέπει επίσης η οδηγία αυτή να είναι τέτοια ώστε να μην ανατραπεί σε μια ενδεχόμενη προσφυγή στο δικαστήριο. Τρίτον, θα πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή η οδηγία κατά την τρέχουσα βουλευτική θητεία, διότι οι προδιαγραφές διαβίωσης για τους παραγωγούς οπωσδήποτε πρέπει να βελτιωθούν και μάλιστα πολύ πριν να γίνει η Κοινοβούλιο να διαχειριστεί. Αυτό που επίσης όμως είναι σημαντικό είναι το να μπορέσουμε να διατηρήσουμε το εισόδημα των γεωργών σε ένα αξιοπρεπές επίπεδο. Είναι ανάγκη να συνεχίσουμε λοιπόν τις διαπραγματεύσεις και να ξεκαθαρίσουμε το σημείο και της δικαιοσύνης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό βρίσκεται στην ουσία της δουλειάς. Όπως είπε και η Μαγκίνες, είναι ανάγκη να δώσουμε προτεραιότητα στην ποιότητα του κειμένου αυτό. Να δούμε αν υπάρχουν ε, λανθάνοντα σημεία που θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε. Είναι πολύ σημαντικό, ούτως ώστε και τη διατήρηση του γεωργικού τομέα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. μου.